Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε. Γιατί ήδη έχουμε καθυστέρηση. Okay, can I ask everybody Καθίστε. Καθίστε παρακαλώ, έχει θέσεις πίσω. Okay, first of all, I would like to welcome everybody back. Σας καλωσορίζω για την επιστροφή σας στο Κοινοβούλιο το νέο αυτό έτος. Ελπίζω να περάσατε καλές διακοπές και το 11 να πάει πολύ καλά. Λέω να αρχίσουμε αμέσως γιατί έχουμε πολύ φορτωμένη μέση διάταξη και μειωμένο χρόνο. Το 11 θα είμαι ακόμη αυστηρότερη από ότι το 10. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να εγκρίνετε τη σύσταση των συντονιστών και συντονιστριών να οριστούν οι επόμενοι εισηγητές. Βιμ για την ενιαία αγορά, την κυρία Φραντσέσκα Κέλλερ για την κατάσταση της κυρίας Φλότρος, εισηγήτριας στη γνωμοδότηση για τις μεταναστευτικές ροές που προκύπτουν από την αστάθεια. Αν δεν έχει κανεί αντίρρηση, όχι. Ε, τότε εγκρίνονται οι προτάσεις αυτές των συντονιστών και συντονιστριών. Επίσης, οι συντονιστές και συντονίστριες που συναντούνται αύριο θα συζητήσουν και πώς πρέπει να χειριστεί η Επιτροπή μας το θέμα του τελευταίου γκρικού νομοσχεδίου για τα μέσα ενημέρωσης και προτείνεται να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής ΕΛΕΦ την επόμενη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Αν το εγκρίνουν οι συντονιστές και οι συντονίστριες θα σας το πω αμέσως. Έχει επίσης προσθεθεί μια συνεδρίαση στις 28 Φεβρουαρίου Τρίτη, 3 με 6.30. έγκριση των πρακτικών δύο τελευταίων συναντήσεων ΕΛΕΦ, όχι δύο λέει αλλά τρεις είναι 4 Μαρτίου, Ιούνιο και Σεπτέμβριο. Μήπως κανείς ή καμία έχει κανένα σχόλιο για τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών. Όχι. Να τότε καλά. Εγκρίνονται. Πάμε τώρα στο σημείο 4 σεξουαλική κατάχρηση παιδών και παιδική πορνογραφία. Θα σας θυμίσω πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Αγγελίλη ότι η κατάσταση των πλογιών έχει λήξει και ότι θα γίνει μία πρώτη ψηφοφορία στις 3 Φεβρουαρίου χωρίς καθέστερο καθυστέρηση. Λοιπόν, δίνω λόγο στην κυρία Αγγελίλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω το σχέδιο έκθεση στην συντομία. Πρόκειται για μία πρόταση που προσπάθησα να εκπονήσω έχοντας κατά νου και τις ενδείξεις ε, των ε, σκιώδων εισηγητών με τους οποίους συναντήθηκα από Λάκης. Στην πρόταση αυτή έχουμε ως σημείο αναφοράς ε, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και επομένως παρά το ότι αυτή η σύμβαση δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη θέλαμε παρόλα αυτά να θεωρήσουμε σε ένα σημείο αναφοράς. Ο στόχος της πρότασης είναι να επικαιροποιήσει την νομοθεσία στο θέμα της καταπολέμησης και της πρόληψης της σεξουαλικής κατοποίησης των παιδιών και της εκμετάλλευσης των παιδιών έχοντας ε, κατά νου και τις τεχνολογικές εξελίξεις ε, του τελευταίων ετών. Οι κύριοι στόχοι ο κύριος στόχος μάλλον ε, είναι να θεσπιστούν ποινές ε, πιο αποτελεσματικές ε, και κατάλληλες, να προβλεφθούν επίσης νέα είδη εγκλήματος όπως είναι το grooming δηλαδή προσέγγιση ενηλίκων με σκοπό την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, αλλά και να έχουμε και μία σειρά μέσων για την πρόληψη αυτών των αδικημάτων, έτσι ώστε να δράσουμε προκειμένου οι και να μην είναι θύματα εκμετάλλευσης και βίας. Επίσης, ε, έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή στην αρρωγή που δίνεται στα θύματα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις ε, έρευνες και τις διαδικασίες και τις δίκες ε, για να αποφύγουμε το φαινόμενο της ε, διτής θυματοποίησης. Της δευτερογενούς θυματοποίησης. Έχουμε και το θέμα των επιβαρυντικών περιστάσεων όταν συντρέχουν τέτοιες περιστάσεις, όταν ε, τα εγκλήματα γίνονται στο εσωτερικό της οικογένειας ή όταν διαπράττονται από ένα άτομο που κατέχει δεσπόζουσα θέση, κυρίαρχη θέση ή ασκεί εξουσία απέναντι στον ανήλικο που είναι το θύμα των πράξεων αυτών και υπάρχουν και πιο αυστηρές ποινές στην περίπτωση που το θύμα είναι άτομο με ειδικέ ανάγκες. Σε ό,τι αφορά επίσης τη διάδοση online επιγραμμική διάδοση παιδοπορκοναφικού υλικού. Ο κύριο στόχος ε, είναι να θέσουμε σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψουμε τα περιεχόμενα στην πηγή. Σε σχέση με την προτεραιότητα αυτή, η φραγή μπορεί να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό και χρήσιμο εργαλείο, η φραγή των ιστοσελίδων, κυρίως στην ε, περίπτωση που δεν είναι δυνατό αμέσως να εξαλείψουμε, να καταργήσουμε στην πηγή όλα τα περιεχόμενα τέτοιου υλικού. Όμως ο στόχος είναι στην πηγή να εξαλείψουμε αυτό το παράνομο περιεχόμενο. Θα περιοριστώ εδώ. Ο στόχος είναι, όπως και εσείς είπατε, να εγκριθεί αυτό το έργο σε λογικό χρόνο προσπαθώντας επίσης να εργαστούμε σε συνέργεια, σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να έχουμε ένα κείμενο με το οποίο θα συμφωνούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και για τη συντομία σας. Ήδη έχω οκτώ αιτήσει για το λόγο. Θα δώσω αρχικά σε όλους δύο λεπτά χρόνο, τώρα 10-11 μάλλον άτομα ζητούν το λόγο. Κάποιος άλλος Θέλει να προσθεθεί. Γιατί είπα ότι βλέπω όλοι όσοι είναι εδώ σχεδόν ζήτησαν το λόγο. Όλοι θα έχουν δύο λεπτά αυστηρά. Ξεκινήσουμε με την κυρία Στρίφλερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Τζελίνη για την εξαιρετική δουλειά της. Ε, εγώ συμφωνώ ε, με όσα είπε η συγγήτρια. Είπατε ότι θέλετε εδώ στο στόχο, να, ε, ο στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά στις δικαστικές διαδικασίες. Πολλές φορές μέσα στην οικογένεια γίνονται τα εγκλήματα και τα παιδιά πολλές φορές δεν κατανοούν το βεληνικές τις δράσεις τις οποίες είναι θύματα. θα πρέπει πρέπει να καλυψούμε τα παιδιά κάθε ηλικία. Θέλω να υπογραμμίσω ότι σε σχέση με το grooming και η διαφορά του σε αυτή την εκδόση είναι ένα καινοτόμο, πολύ θετικό στοιχείο και πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε όλους τους ανηλίκους και τους γονείς για τον ενδυνάμει επικίνδυνο χαρακτήρα που μπορεί να έχουν οι επικοινωνίες στο ίντερνετ και ποια αντίδραση θα πρέπει να έχουν, πια αντανακλαστικά για να μπορούν να σωθούν. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο να ενημερώσουμε και τους γονείς και τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σίπερ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, η οποία πραγματικά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στον τομέα τη πρόληψη και στην αναφορά στην ε, εκμετάλλευση που γίνεται σε οικογενειακό επίπεδο και που τονίζει ιδιαίτερα τη βοήθεια για τα θύματα mm. κάθαρα και μέχρι την ουσία τους γιατί ξέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν ε, καθυστερημένες επιπτώσεις αυτών των κακοποιήσεων και εκμεταλλεύσεων και είναι σωστό να αναφέρεται στην οδηγία. Θα ήθελα ταυτόχρονα όμως να πιστήσω την προσοχή της εισηγήτριας σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στο θέμα της αύξησης των κυρώσεων και σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν μάλιστα για να ξέρουμε γιατί γίνεται αυτό που γίνεται. Μετά υπάρχει στην τροπολογία 28 ένας περιορισμός, δηλαδή η Κομισιόν πρότεινε οι δράστες να αποκλείονται από οποιασδήποτε δραστηριότητες τους φέρνουν σε συνεχή επαφή με παιδιά στην τροπολογία αναφέρεται αυτός ο αποκλεισμό θα πρέπει να ισχύει μόνο για επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτός είναι ο περιορισμός λοιπόν και δεν ξέρω. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Μετά υπάρχει μια νέα παράγραφος, παράγραφος 36, όπου διευκρινίστε για άλλη μια φορά ότι αν είναι δυνατόν δεν θα πρέπει η εξέταση των ε, παιδιών θυμάτων να γίνεται παρουσία του δράστη. Αυτό ε, θα πρέπει να δούμε, ε, θα πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά κατά πόσο το παιδί θα πρέπει πραγματικά να εξαρτηθεί παρουσία του δράστη. Η Κομισιόν βλέπω ότι κάνει διαφορετική αξιολόγηση του κατά πόσο θα διαγραφεί ή θα μπλοκαριστεί αυτό όμως δεν προβλέπεται δεσμευτικά και δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνατότητα τροποποίησης και εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ παρακαλώ μην ξεχνάτε το ρολόι. Δεν θέλω να είμαι κακιά, αλλά δεν έχουμε σαΐ χρόνο. Ρέβα την επόμενη, επόμενη συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, διευκρινίσαμε νομίζω απόλυτα ότι σε πολλά σημεία Η πρόταση δεν είναι τέλεια. Πολλά από τα σημεία θα αναφερθούν βέβαια. Εγώ θα περιοριστώ σε ένα θέμα. Τη συζήτηση για το, ε, την απόκρυψη ιστοσελίδων. Και ε, αυτό δεν θα πρέπει να ε, λέμε ότι είναι θέμα που αφήνεται στα κράτη-μέλη λέγεται τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να υιοθετήσουν μέτρα για τη φραγή αυτών των ιστοσελίδων. Εμείς τα λέγαμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να το κάνουν χωρίς να αναφέρουμε το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να δράσουν. Θα θέλω λοιπόν η θέση του Κοινοβουλίου να είναι πιο σαφής ότι αυτή η φραγή δεν είναι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε εμείς θέλουμε να πετύχουμε την διαγραφή αυτού του υλικού από το διαδίκτυο. Και βλέπουμε κάποιες προτάσεις οι δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα. Θα ήθελα να πω να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακόμα στοιχεία ότι η διαγραφή δεν είναι ε, καλή, δεν λειτουργεί. δεν ξέρω κατά πόσον κατελήφθησαν προσπάθειες να υπάρξει συνεργασία με εκείνες τις χώρες που δεν συνεργάζονται για το θέμα της διαγραφής. Εφόσον δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, η φραγή δεν είναι αυτό που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στην οδηγία. Και αν υπάρχει αναφορά στην φραγή δεν θα μπορεί να γίνεται εξοδικαστική γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο με τις ε, ε, διατάξεις ε, που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελευταία λέω ότι υπάρχουν ενώ ένομα μέσα και αν δεν τα ακολουθήσουμε για την φραγή δεν θα είμαστε ευθυγραμμισμένοι με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. We have until quarter to four. Κοιτάξτε, μέχρι τις 4 παρατέταρτο έχουμε χρόνο. Λοιπόν, η κυρία Βίξτρομ έχει το λόγο και μετά η κυρία Ένστ. Σας κατευχαριστώ Πρόεδρε καθώς και τον εισηγητή για την ωραία του έκθεση, την ωραία της έκθεση εισηγητή. Και μου άρεσαν πολύ αυτά που είπε ο τελευταίος ομιλητής αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κύριο θέμα είναι τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν όποτε υπάρχει ο φόβος ότι κάτι μπορεί να βλάψει ένα παιδί να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το κύριο πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν πρέπει να επιβάλλουμε σε όλες τις χώρες μέλη φραγές. Να λέμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποσβήσουν, να σβήσουν αυτές τις ιστοσελίδες και ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη φραγή ως συμπληρωματικό μέσο όποτε δεν μπορεί να επιτευχθεί η απαλήφη. Όταν ο εξυπηρετητής βρίσκεται στις Ηνωμένε Πολιτείες ή στην Πολιτείε η σελίδα. Αλλά όχι όταν βρίσκεται σε αλλού στα λεγόμενα phishing sites. Εκεί δεν μπορούν να σβηστούν οι ιστοσελίδες αποτελεσματικά και γρήγορα, ενώ πρόκειται για τρομερό έγκλημα που πρέπει να καταπολεμηθεί με κάθε τρόπο. Επίσης νομίζω ότι πρέπει να προσέχουμε τη διατύπωση. Πολλά κράτη-μέλη έχουν δικά τους συστήματα, έχουν δικά τους συστήματα για τις ποινές που επιβάλλονται. Ξέρω ότι υπάρχουν μερικοί άρρωστοι άνθρωποι που χρειάζονται μάλλον θεραπεία παρά τιμωρία και φυλάκιση και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η εισηγήτρια επίση λέει ότι οποιοδήποτε καταδικάστηκε για έγκλημα σχετικό με παιδιά δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να ασκήσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με παιδες. Αλλά αυτό είναι πολύ ευρύ. Το θέμα είναι σημαντικό και πρέπει να επανέλθουμε πολλές φορές. Ευχαριστώ. Κυρία Έρνστ, σας ευχαριστώ. Και μετά ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το θέμα της πρόληψης. Ότι η πρόληψη δηλαδή θα πρέπει να αποκτήσει εδώ μεγαλύτερη σημασία και πολύ πιο εδαφροποιημένα γίνεται αυτό στην έκθεση. Είναι πάρα πολύ καλό και το υποστηρίζουμε. Το επόμενο είναι ότι έχω παρόμοιε ερωτήσει όπω και η κυρία είπε. Γιατί αυξήθηκε το επίπεδο των κυρώσεων, ε, υπήρχε κάποιο κίνητρο, γιατί υπάρχει παντού μια αύξηση ενό έτου. Γιατί. Και εκείνο που θα ήθελα να εκφράσω είναι το θέμα της ε, ε, διαγραφής και της φραγής. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει ξεκάθαρα να πούμε ότι θα θέλουμε να υπάρχει η διαγραφή. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Να δούμε παντού τις διατυπώσεις που αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου σαφής. Γιατί οι δυνατότητες φραγής που προβλέπονται δεν είναι και δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ας πούμε για την προειδοποίηση των δραστών. Και αυτό δεν θα πρέπει να το δεχτούμε. Παρακαλώ λοιπόν αυτό το θέμα να ξανεξαρτηθεί σαφώς και να διατυπωθεί διαφορετικά από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και θα ήθελα να ε, παρακαλώ τη συζητήτρια να λάβει υπόψη και τις φωνές που ακούστηκαν από τις μη κυβερνικές οργανώσεις, από οργανώσεις θυμάτων που ήρθαν σε επαφή με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να βελτιωθεί, το σημείο. Αυτό σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ο κύριος και μετά η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Αντζελίνη που εκπώνησε τόσο γρήγορα την έκθεσή τη. Πολύ καλή δουλειά έχει κάνει στην εισαγωγή ορισμένων προληπτικών μέτρων ε, που έλειπαν εντελώς από την αρχική πρόταση της Κομισιόν, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόνται περισσότερα για να ε, δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την πενικοποίηση ε, του δράστη. Πιστεύω ότι τα προληπτικά μέτρα είναι αδύναμα και γενικά και εμφανίζονται μόνο στα εκτιμώντες επίση η προστασία που παρέχεται στα θύματα σχετίζεται πάρα πολύ στενά με τι ε, ποινικέ διαδικασίε. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ θεωρώ ότι αυτή η υποστήριξη δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη συμφωνία για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια τη δίκη και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερε συνθήκε του παιδιού και για την τελευταία πρόταση τη διαγραφή υφραγή των η δική μα ομάδα. Φυσικά συμφωνεί με τα περισσότερα που είπαν οι συνάδελφοι εδώ για την διαγραφή. σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χίρς και κατόπιν ε, κυρία Κεντρισούτα. Ähm, Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Συζητήτρια των Φιλευθέρων στην Επιτροπή Πολιτισμού. Θα χαίρομαι πολύ που συζητιέται το θέμα αυτό και στην Επιτροπή Ελευθεριών και θα ήθελα να ε, συγχαρώ την συγγήτρια για τα προεπτικά μέτρα που ανάφερε και εμείς είχαμε υποβάλει κάποιες σχετικές προτάσεις. Μου φαίνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ενημέρωση για να μην φτάνουμε να ε, διαπράττονται αυτές οι πράξεις. Εκτός αυτού το θέμα της αύξησης του επίπεδου των κυρώσεων θα πρέπει να δούμε κατά πόσον είναι λογικό να εγκαταλείψουμε την συστηματική προσέγγιση των κρατών μελών γιατί αυτό ίσως στρεβλώνει και τη σχέση αυτών των κυρώσεων με κυρώσεις για άλλα ε, ε, παραπτώματα ή <coughs> δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι εμείς στην Επιτροπή Πολιτισμικών Θεμάτων έχουμε μια πολύ καλή και ακριβή διατύπωση ε, για την παράγραφο 21 ότι η διαγραφή είναι το πιο σημαντικό και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια γεννή αυτό. Και αυτό δεν είναι ιδεολογική συζήτηση, είναι θέμα της προστασίας των θυμάτων. Γιατί άμα το κοιτάξουμε τα πράγματα από προοπτική των θυμάτων, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τα άτομα αυτά είναι αυτές οι εικόνες να εξαφανιστούν από το διαδίκτυο και να μην μπορεί κανένας πια να έχει πρόσβαση σε αυτές. Από την προοπτική δηλαδή της προστασίας των θυμάτων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαγράψουμε και αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να το πετύχουμε αυτό να έχουμε κατά νου Αλλά θα πρέπει πάλι να πούμε ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιο τυχαίος αλλά θα πρέπει να γίνεται αυτό κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλιώς ε, δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε και θα αρχίσουν οι τι πρέπει να διαγραφεί, τι δεν πρέπει να διαγραφεί κλπ. Αλλά θα πρέπει να είναι σαφέ. Πρώτα διαγραφή και μετά φυλακή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε άλλους τομείς υπάρχει ακριβώς καλή συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και θα μπορεί να γίνει το ίδιο και εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπλεγεβισούτα και μετά ο κύριο Πάσκορ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, πολύ καλή έκθεση και θέλω να υποστηρίξω την πρόταση ότι θα πρέπει να έχουμε συμπληρωματικές συζητήσεις, ε, μάλλον θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις για αυτή την οδηγία το συντομότερο. Γιατί πρέπει να οδηγηθούμε στην έγκριση αυτή της οδηγίας. Θέλω να τονίσω ότι δεν έχουμε επαρκή στατιστικά στοιχεία για τα κράτη-μέλη σε σχέση με την κακοποίηση των παιδιών και για το πορνογραφικό υλικό που απεικονίζει παιδιά, κυρίως όταν μιλάμε για περιπτώσεις εντός οικογενειών. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό το θέμα στην έκθεση. βάση της πρακτικής εμπειρίας θα ήθελα να πω ότι βλέπουμε να υπάρχει έλλειψη ειδικών, ε, όπως ψυχολόγων και άλλων ειδικών, που θα έχουν εκπαιδευτεί για να εργαστούν στον τομέα αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να προβούν στην εκπαίδευση τέτοιων εμπειρογνωμόνων που θα ξέρουν πώς να χειριστούν τα θύματα. Τώρα για το άρθρο 21, για τη διαγραφή ε, των ιστοσελίδων, αυτών που έχουν υλικό και είμαι υπέρ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχασε ένα τμήμα της παρέμβασής σας, κυρία Μπόσκουρτ, και κατόπιν κύριος Σμίλντερ. Ehm, eh, ehm, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την συγκέντρια για την πάρα πολύ καλή και σημαντική εργασία που επετέλεσε. Το θέμα που θα ήθελα να εξετάσω είναι το θέμα του μέχρι πότε θα μπορούμε πραγματικά να θεωρήσουμε ότι μπορούμε να διώξουμε κάποιον που την τελευταία στιγμή αποδεχτεί ότι ήταν δράστης στο παρελθόν. Αυτό. Πότε δηλαδή παραγράφονται αυτά τα εγκλήματα. Το δεύτερον, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το θέμα ότι αυτή η δράση δεν θα επιτρέπεται στην επαγγελματική σου ζωή να έχουμε επαφή με παιδιά ούτε επαγγελματικά ούτε σε εθελοντική βάση. Και αυτό θα ήταν κάτι πράγμα παρακαλώ που θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Ευχαριστώ. Προσεγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μιλτερ. και ο κύριος Φως τελευταίος και μετά εγώ. Uh, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και στην εισηγήτρια. Προέρχομαι και εγώ από την ίδια χώρα με την παρέμβαση της κυρίας Βόρστ, δηλαδή ότι αν ε, θέλει κάποιος ε, να εργαστεί σε κάποιον οίκο παιδιών, τότε θα πρέπει να λαμβάνει ε, το κατάλληλο έγγραφο από την αστυνομία. Στην τελευταία περίπτωση που είχαμε στις κατοχώρες, αυτό το λαμβάνουμε από τις εθνικές αρχές. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα γνωρίζουμε τι έχει γίνει με το άτομο αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένα μητρό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ανταλλάζουμε πληροφορίες για τις καταδίκες έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος ε, που θα έχει ποινικό μητρό ε, για τέτοιου είδους εγκλήματα να μην μπορεί να προσληφθεί σε χώρους όπου υπάρχουν παιδιά. Και εγώ θέλω να κάνω μια τροπολογία προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Κύριε Βος. Σας ευχαριστώ. Εάν θέλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη το θέμα της καταπολέμησης της θερικής ε, πορνογραφίας, δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε από το θέμα της φραγής των ε, ιστοσελίδων. Τώρα, θα πρέπει να πούμε φραγή μέχρι να υπάρχει διαγραφή ή καταρχήν διαγραφή και αν δεν καταφέρουμε τη διαγραφή να υπάρχει φραγή. Θα πρέπει να το δούμε αυτό και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι σελίδες μπορούν να ε, είναι διαθέσιμες μέχρι να διαγραφούν και θα υπάρξει πάντα έτσι μια δυνατότητα παρέμβαση στην ε, δημόσια τάξη. Mm. Και γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της φραγής. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή να δούμε πώς θα το εφαρμόσουμε και πώς θα πετύχουμε να καταστεί αυτό υποχρέωση και όχι μια δυνατότητα των κρατών μελών. Εγώ λοιπόν θα ήθελα καταρχήν φραγή ξεκάθαρα και μετά θα δούμε πώς θα γίνει αυτό στις λεπτομέρειες του. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει, θα ήθελα να πω και εγώ δύο πράγματα. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία της για να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να τονιστεί περισσότερο το γεγονός ότι παρόλο που αυτά που δημιούργονται στο διαδίκτυο είναι φοβερά λόγω το θέμα του θέματος της διάδοσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνουν χώρα στα, στις στα σχολεία, από άτομα που τα παιδιά τα εμπιστεύονται. Θα ήθελα λοιπόν να τονιστεί περισσότερο το θέμα γι' αυτό της πρόληψης και των κυρώσεων επίσης προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερον, φραγή η διαγραφή, καλά κινηθήκατε νομίζω που είπατε ότι καλύτερα ήταν να είπε διαγραφή και τονίσετε λιγότερο τη φραγή. Είπανε και άλλοι συνάδελφοι ότι παραμένουν πολλά ερωτηματικά για τη φραγή και θα ήθελα εγώ να στραφώ προς την Κομισιόν άμεσα. Γιατί εγώ έχω αποβάλει μία ε, κοινοβουλευτική υπερώτηση αναρωτιόμουν γιατί μέσα στα πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας η ίδια η Κομισιόν α, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η φραγή είναι τελείως αναποτελεσματική. Λοιπόν, εάν θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, γιατί θεωρεί η Κομισιόν ότι είναι το ίδιο μέτρο αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της παιδικής τρομοκρατίας. Γιατί θέλει να το χρησιμοποιήσει σε αυτή την περίπτωση της αποφύγησης κακοποίησης των παιδιών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Μπορατίτσκι και τον κύριο Λούζο Ιρεάτη της Κομισιόν να σχολιάσουν. Δεν ξέρω ποιος από τους δυο τους. Ευχαριστώ πολύ που μας κάνετε λόγο. Γιάκο λέγομαι. Καταρχήν θέλω να σας ε, ευχαριστήσω για το ότι εξετάσατε εις βάθος την πρότασή μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Αντζελίνη, όπως ε, και τους σκιώδους συζήτητες σε άλλες επιτροπές που συζήτησαν το σχέδιο του κειμένου. Καλωσορίζουμε μία σειρά από τροπολογίες και προτάσεις που γενικά ενδυναμώνουν το μήνυμα και το στόχο της οδηγίας. Και θέλω να συμφωνήσω με όσα είπατε, Πρόεδρε, ότι η οδηγία έχει να κάνει με πολλά θέματα που ξεπερνούν το διαδίκτυο. Και η αξία αυτής της νομοθεσίας είναι ότι είναι ένα συνολικό εργαλείο που θέλει να προστατεύσει τα παιδιά κατά τη σεξουαλική κακοποίηση που λαμβάνει χώρα στην πραγματική ζωή. Να υπενθυμίσω ότι όταν ε, μιλάμε για παιδική πορνογραφία και διάδοση αυτού του υλικού στο διαδίκτυο, μιλάμε και για μία κακοποίηση που έλαβε χώρα κάποια στιγμή στην πραγματική ζωή. Πολλά υπόθηκαν για τη φραγή. Η Κομισιόν διατηρεί τη θέση της πράγματι ότι η φραγή είναι σημαντική δραστηριότητα που λαμβάνεται από τις διοκτικές αρχές και έχει καταλήγει στην αφαίρεση του παρανομηλικού. Βλέπουμε σημαντική διαφορά μεταξύ της τρομοκρατίας ε, γιατί εκεί στοχεύουμε σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων και μεταξύ ε, φραγή των σελίδων παιδικής πορνογραφίας. Όταν μιλάμε για ε, παρεμπόδιση ατόμων σε τέτοιο υλικό και παρεμποδίζουμε όχι μόνο τους παιδόφιλους αλλά και γενικά το κοινό. Πολλά επιχειρήματα ακούστηκαν κατά της φραγής. Τι παρατηρήσαμε εμείς, ότι πράγματι αυτό θεωρείται ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της παιδικής ε, παρνογραφίας σε αρκετές χώρες, ε, με το σχάρι Ιταλία, Σουηδία, Ενωμένο Βασίλειο. Και αυτό σχετίζεται κυρίως με το γεγονός ότι δυστυχώς παρά πολλών προσπαθειών η διαγραφή δεν γίνεται αμέσως και καθώ οι περισσότερε του σελίδε είναι εκτό δικαιοδοσίας τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η διαδικασία χρειάζεται χρόνο. Να υπενθυμίσω τι πρόσφατε συζητήσει που έλαβαν χώρα στη Γερμανία, όπου η Criminal Act ανέφερε τις δραστηριότητές της ε, σε μια κρόαση που έλαβε χώρα στις 25 Οκτωβρίου στο Bundestag, στο Κοινοβουλίο όταν ε, οι ε, αστυνομικοί είπαν ότι παρά τις ε, προσπάθειες που κατεβαλάν το 45% των σελίδων που φιλοξενούνται στο εξωτερικό εξακολουθούν να είναι online και δεν έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση. Έχουμε αρκετά παραδείγματα γιατί δεν λειτουργεί αμέσως η διαγραφή. Δεν θέλουμε βέβαια τώρα να επιμηκύνουμε τη συζήτηση εδώ για το phishing. Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά. Έχουμε εδώ, ε, παραδείγματος χάρη, ε, έναν οργανισμό που μπορεί να λάβει όλα τα μέτρα ε, για ε, να γίνει, εφαρμοστούν τα μέτρα, ενώ στην περίπτωση της παιδικής πορνογραφίας έχουμε ένα παιδί και ένας πολίτης οφείλει, ε, παραδείγματος χάρη, να καταγγείλει την ε, απάτη, όμως στην περίπτωση που έχουμε παιδική πορνογραφία ε, τότε δημιουργούνται κάποιες υποψίες, δηλαδή θα αναρωτηθούμε εσύ ως πολίτης έπεσες πάνω σε αυτό το υλικό. Και καθώς είναι παράνομη η φύση αυτού του υλικού, ο ίδιος ο χειρισμός μπορεί ε, να θεωρηθεί αδίκημα. Πάντως εκτιμούμε τις βάθο συζητήσει ε, που γίνονται στο Κοινοβούλιο. Μάλιστα εμείς καλέσαμε και τους ε, σκιώδεις εισηγητέ και την εισηγήτρια σε επισκέψεις, μελέτες που οργανώθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το κέντρο που ασχολείται με την εκμετάλλευση, τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και έχει ως στόχο να προστατεύει τα παιδιά κατά της σεξουαλικής κακοποίησης, ασχολείται και με την έρευνα και με την προστασία των θυμάτων, όπως ε, και τη φραγή και τη διαγραφή των σελίδων την ε, Τετάρτη λαμβάνει η χώρα αυτή η δραστηριότητα. Υπάρχουν λοιπόν ε, και άλλοι ευρωβουλευτέ ή βοηθοί των βουλευτών που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτέ τι επισκέψει, ε, φυσικά και του προσκαλούμε εκ μέρου αυτή τη αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου που συνδιοργανώνει μαζί μα αυτή την επίσκεψη. Ένα ακόμη συγκεκριμένο ζήτημα, Πρόεδρο. Μπορείτε να είστε πιο σύντομο, ναι, δεν θα αναφερθώ σε άλλο ουσιαστικά σε μια ο να αναφερθώ και στο παραδείγμα των ε, κατοχωρών. Ε, φαίνεται ότι υπάρχουν ε, αποτελεσματικές δραστηριότητες προς αυτήν την κατεύθυνση και πάλι η Κομισιόν θέλει να ε, σας αναφέρει ότι δεν έχουμε στην αρχική πρόταση περιορισμό μόνο στις επαγγελματικέ δραστηριότητες. Επίσης, ε, μαζί με την ε, Προεδρία συζητήσαμε αυτή την πρόταση. Πριν τα τέλη του έτους ολοκληρώσαμε το έργο με το Κοινοβούλιο για την Οδηγία για την Εμπορία Ανθρώπων, ε, που ήταν το πρώτο μέσο ποινική φύσεως μετά τη συνθήκη της Λισαφώνης. Και βλέπω εδώ και την κυρία Μπάουρ που αντιδρά. Και θέλουμε να έχουμε μια ταχύ διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν συνοψίσει η συγκήτρια θα ήθελα να πω ότι οι διαφορές που σημειώσατε μεταξύ καταπολέμησης τρομοκρατικών ιστοσελίδων και παιδεραστικών αυτών ε, είναι μικρή. Δηλαδή το πιο σημαντικό που είπατε είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος για να καταπολεμηθούν και τα δύο είδη ιστοσελίδας η αστυνομία για να αναφέρει καν και μόνο την ύπαρξη αυτής της ιστοσελίδας χρειάζεται να ακολουθήσει μια πολύ μακροσκελή διαδικασία, αλλά αυτό δεν είναι θέμα τεχνικό. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε. Να μην μπλοκαριστούν όλα επειδή δεν έχουμε σωστά βάλει τις προτεραιότητες μας. Κυρία Αγγελίλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους καταρχήν για όλες τις παρατηρήσεις τους και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνθεση ξεκινώντας από ένα επιχείρημα που νομίζω ότι αναφέρθηκε από όλους. Δηλαδή, η προτεραιότητα της διαγραφής των ε, παιδοπορνογραφικών στο σελίδων online ή τη φραγή. Εμείς ε, ε, Είχαμε πάρα πολλές ε, μαρτυρίες ε, και αναφέρθηκαν πάρα πολλές πρακτικές εμπειρίες, κυρίως από κάποια κράτη-μέλη, που έχουν να κάνουν ακριβώς με τη διαγραφή των ε, πορνογραφικών ιστοσελίδων. Εγώ προσπάθησα στο κείμενο να είμαι, να σαφής, αλλά φυσικά μπορώ να κάνω και επιπλέον διορθώσεις. Ο κύριος στόχος η προτεραιότητα είναι η διαγραφή στην πηγή των παράνομων ε, και επικίνδυνων περιεχομένων. Αυτός είναι ο μόνος στόχος. Όμως η φραγή μπορεί να είναι χρήσιμη και συμπληρωματική σε δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή η διαγραφή της ιστοσελίδας, ε, γιατί μπορεί ο σερβερ να βρίσκεται εκτός της ευρωπαϊκής κοινότητας και ίσως είναι δύσκολο να φτάσουμε στην πηγή. Αλλά ακόμη και όταν είναι δυνατή η διαγραφή, αλλά χρειάζεται χρόνος. Μπορεί να χρειαστεί μία μέρα, μία εβδομάδα ή ακόμη και 6 ώρες. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη και το επενθύμησε η Κομισιόν ε, η ΣΕΟΠΑΛΑ και η ε, αστυνομία, ταχυδρομική αστυνομία τη Ιταλίας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε λίγα λεπτά μπορούν να παρέμβουν και να μπλοκάρουν την εικόνα για να έχουν το χρόνο στη διαθεσή του για να διαγράψουν το περιεχόμενο. Αν χρησιμοποιηθεί λοιπόν η φραγή για την άμεση παρέμβαση, για την άμεση επέμβαση, εγώ νομίζω ότι μπορεί να αποτελεί η φραγή συμπληρωματικό εργαλείο. Αλλά το επιθυμίζω, η διαγραφή του περιεχομένου είναι ο στόχο. Ήθελα να είμαι λοιπόν απόλυτα σαφής για το θέμα αυτό. Κατόπιν. Δέχτηκα όλες τις παρατηρήσεις ε, που αφορούν την πρόληψη της κακοποίησης, ε, την ενημέρωση που πρέπει να δίνεται όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους, αλλά και στους ε, εκπαιδευτικούς και στους όσους ασχολούνται με παιδιά. Και επίση ε, και την κατάρτιση του προσωπικού. Η κατάρτιση μπορεί να είναι κατάρτιση του προσωπικού στα σχολεία. ή των αστυνομικών όπως και όσων διαδραματίζουν ε, ένα ρόλο στη δικαστική διαδικασία. Είναι απαραίτητη η παροχή ενημέρωσης. Συμφωνώ για το ότι πολλές ε, κακοποίησεις συμβαίνουν στο εσωτερικό της οικογένειας. Μπορούν ε, να γίνουν και στο σχολείο. Και σε αυτό, βλέπουμε λοιπόν ότι συμβαίνουν σε πάρα πολλές προστατευμένες εισαγωγικά καταστάσεις. Εκεί πρέπει να δράσουμε αποφασιστικά γιατί κάποιος ε, εκμεταλλεύεται μία θέση εξουσίας ή συγγένειας για να προβεί σε κακοποίηση. Και αυτό είναι τρομερό. Κατόπιν. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ποια από τις συναδέλφους αναφέρθηκε. Μάλιστα. Η κυρία Σίπελ μου ζήτησε κάτι για την τροπολογία 28 Η τροπολογία 28. Αναφέρεται στην ανταλλαγή ενημέρωσης μεταξύ των κρατών μελών και των ποινικών μητρώων, έτσι ώστε να αποφύγουμε άτομα που έχουν ε, καταδικαστεί για σεξουαλικά δικήματα να μην μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητες σε επαφή με παιδιά. Εγώ περιορίστηκα στο να αναφερθώ εδώ στις επαγγελματικές δραστηριότητες. Αυτό το έκανα γιατί κατά την άποψή μου ήταν πολύ γενική η διατύπωση της Κομισιόν. Όμως ε, πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε ένα συμβιβασμό έτσι ώστε να διευκρινιστεί καλύτερα το ζήτημα γιατί διαφορετικά νομίζω ότι το Συμβούλιο δύσκολα θα μπορούσε να δεκτεί μια τόσο γενική πρόταση, αλλά συμφωνώ ότι θα έπρεπε να διευκρινίσουμε καλύτερα τα θέματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι ελάχιστε ποινέ και την αύξησή του, αρκετοί συνάδελφοι με ρώτησαν γιατί πρώτη αύξηση κατά ένα χρόνο τη ελάχιστη ποινή. Το έκανα γιατί υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που ε, ζήτησαν να υπάρχει αύξηση, αναφέρονται μάλλον αρκετά κρατημέλη σε σχέση με την αύξηση κατά ένα έτος αυτής της ποινής, της ελάχιστης ποινής. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να ξανασυντηθούμε με τους και οδησυγητές είτε στο Στρασβούργο είτε μετά από την προθεσμία λήξης για την κατάσταση τροπολογιών για να προτιμάτε στη δεύτερη περίπτωση θα στείλω ένα email και βάσει τη και των δικών σας απόψεων. Θα προσπαθήσουμε να συναντηθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα έργο με το οποίο θα συμφωνούν οι περισσότεροι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Αντζελίνη. 28 Ιανουαρίου, το μεσημέρι στις 12 είναι η προθεσμία λήξη για και θα έχουμε ψηφοφορία Φεβρουαρίου. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο, είναι η διαδικασία υποβολή αίτηση για τη χορήγηση τη διαμονή και εργασία. Κυρία Ματιανή, συγκήτρια. Όπω ξέρετε, κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο, το κείμενο απορρίφθηκε στην Ολομέλεια και εστάλει πίσω η έκθεση στη δική μα επιτροπή. Άρθρο 56, παράγραφος 3 του εσωτερικού μας κανονισμού Λέγεται εκεί ότι η αρμόδια επιτροπή σε τέτοια περίπτωση θα αποφασίσει επί τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και προφορικά η γραπτά θα αναφέρει πίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια προθεσμία εντό δύο μηνών. Mm. Έτσι λοιπόν ε, η συγγήτρα και οι σκιώδεις ε, θα πρέπει να υποβάλουν μια πρόταση που να μπορεί να εγκριθεί στην Ολομέλεια. Πράττοντας κάτι τέτοιο πρέπει να λάβουμε υπόψη την, το αίτημα της Επιτροπής Απασχόλησης να συμμετάσχει. Και πάλι στο άρθρο 50 αναφέρεται κάτι τέτοιο, στο άρθρο 50 του κανονισμού. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ ζήτησε από τη Γραμματεία να έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες της Ολομέλειας για το αν ε, υπάρχει κάποιο προηγούμενο που μπορεί να μας καθοδηγήσει στην περίπτωση αυτή. Θα σας ενημερώσουμε για την απάντηση που θα λάβουμε σχετικά με το συγκεκριμένο τρόπο εμπλοκής της Επιτροπής Απασχόλησης. Θα καλέσω τώρα την κυρία Ματιέ πάρει το λόγο και κατόπιν οι συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων παρακαλώ να παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε συμβιβασμό σχετικά γρήγορα. Κυρία Ματιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς η πρόταση όπως έχει τροποποιηθεί απορρίφθηκε στις 14 Δεκεμβρίου και συμβουλευτήκαμε τις υπηρεσίες της Ολομέλειας που μας αποσαφήνισαν ότι δεν υπάρχει προηγούμενο και ότι η Επιτροπή ΕΛΕΦ που είναι η αρμόδια παρά το 50, άρθρο 50 είναι στα χέρια είναι η αρμόδια υπεύθυνη για να ασχοληθεί με αυτό το κείμενο. Επαναπέμφθηκε λοιπόν το κείμενο στην Επιτροπή ΕΛΕΦ και αυτή πρέπει να λύσει το πρόβλημα τους επόμενους δύο μήνες από τη 14 Δεκεμβρίου. Πράγματι λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε τι συμβιβασμό μπορούμε να πετύχουμε και νομίζω ότι για τα σημεία που, όπου σημειώθηκε η μεγαλύτερη διαφωνία μπορούμε ίσως να βρούμε ορισμένους συμβιβασμούς και γι' αυτό θα προτείνω συνάντηση με τους σκιώδεις της ΕΛΕΦ αυτή την εβδομάδα θα δω και σκιώδεις από πολιτικές ομάδες έχω τηλεφωνικό ραντεβού με το γραφείο της κυρίας Μάιλστρομ το απόγευμα σήμερα θα συναντηθώ και με την Προεδρία επίσης αυτή την εβδομάδα για να δω τι, σε τι διατύπωση θα μπορούσαμε να καταλήξουμε που να ικανοποιεί και τις πολιτικές ομάδες και την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Να αυτά μπορώ να σας πω κυρία Πρόεδρε και σε εσά και στους συναδέλφους. Α, άκουσα τις απόψεις τους και θα επανέλθω στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Μήπως πρέπει να μιλήσουν και οι συντονιστές όπως ο κύριος Μπουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχίζω ευχαριστώντας την Βερόνικα Ματιέ, όχι μόνο για την ε, τωρινή της εξήγηση, αλλά και για όλα όσα έχει κάνει για το θέμα αυτό. Είναι κρίμα που τελικά το Δεκέμβριο καταλήξαμε σε απόρριψη αυτό δεν ήταν αναπόφευκτο και είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει εάν οργανωθούμε καλά, στην Επιτροπή μας ιδιαίτερα. Γιατί έχουν υπάρξει παρεξηγήσεις ως προς το θέμα αυτό. Ας μην τις αναφέρω όμως, θα ήθελα αντίθετα να τονίσω πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Συμφωνώ με την κυρία Ματιέ ότι πρόκειται για θέμα που αφού έχει επαναπευθεί σε εμάς εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την επίτευξη συμβιβασμού και λύσης και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει η ΕΛΕΦ κατεπηγόντως να καταλήξει σε μια διατύπωση που να μπορεί να ξαναψηφιστεί στην Ολομέλεια ελπίζοντας να υπάρξει συμφωνία από την πρώτη ανάγνωση. Αυτό το κείμενο βέβαια πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τα αποτελέσματα της ψηφοφο... προηγούμενης ψηφοφορίας ιδιαίτερα ως προς συγκεκριμένες τροπολογίες αν θέλουμε να επανέλθει στην Ολομέλεια και να πετύχει πλειοψηφία. Και έτσι ξαναευχαριστώ την κυρία Βερόνικα Ματιέ αλλά επαναλαμβάνω χρειάζεται ταχύτης γιατί υπάρχει εδώ μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να παραλείψουμε είναι από τα πρώτα νομοθετήματα σε αυτό το σημαντικό τομέα της νόμιμης μετανάστευσης. Ευχαριστούμε. Μωράς. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Ματιού για όλα όσα έχει κάνει. Πάντοτε είναι δύσκολο να βλέπει κανείς ότι δεν υπάρχει τελικά συμφωνία μετά από τόσο πολλή δουλειά. Όπως και ο κύριος Μπουσουτήλ θα ήθελα να πω εξ ονόματος της ομάδας μου ότι θέλουμε οι σκιώδεις να παίξουν όσο πιο επικοδομητικό ρόλο γίνεται μέσα στη διορία αυτή των δύο μηνών για να επιτευχθεί συμβιβασμός. Θα επαναθέσουμε τροπολογίες στην Ολομέλεια και θεωρούμε τα σημεία όπου υπήρξε διαφωνία ως τα σημαντικότερα. Αυτή είναι η βασική θέση που πρέπει να διατηρήσουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις μέσω της κυρίας Ματιού και των σκιωδών, ιδίως τη δική μας, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συνέπεια ως προς την διεύρυνση που ζητιέται από ορισμένου για το πεδίο εφαρμογής του νομοθετήματος. Ως προς το κατά πόσον η Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει και αυτή να παίξει κάποιο ρόλο, εγώ νομίζω δεν είναι θέμα που πρέπει να το δούμε εμείς, αλλά να εξετάσουμε καταρχήν αν υπάρχει προηγούμενο, να το δει η γραμματεία δηλαδή. Εμείς ως Επιτροπή ΕΛΕΦ μόνοι μας Μπορούμε να αναλάβουμε από μόνοι μας όλες τις διαπραγματεύσεις ή πρέπει να συμμετάσχει και η Επιτροπή Απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 50. Αυτό όμως θα το λύσει η γραμματεία, όχι εμείς ως συντονιστές και συντονίστριες. Αλλά ό,τι και να γίνει εμείς στην ομάδα μας θα παίξουμε επικοδομητικό ρόλο στις διαπραγμάτευση με την κυρία Ματιού τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστούμε κυρία Βέμπερ, ο πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ την κυρία Ματιού για τις προσπάθειές της και νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσουμε δύο στοιχεία, το διαδικαστικό από τη μία και την ουσία από την άλλη. Ε, για να χειριστούμε δε την ουσία πρέπει πρώτα να δούμε τη διαδικασία. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει προηγούμενο ακριβώς, αλλά έχει συμβεί κάτι ανάλογο με την περίπτωση αυτή. Ήταν μια επιτροπή αρμόδια για το χειρισμό ενός θέματος, Ήταν λοιπόν μία και τώρα ήταν δύο μάλλον και τώρα μόνο η ΛΥΜΠΕ, η ΕΛΕΦ πρέπει να είναι αρμόδια. Η Επιτροπή Απασχόλησης έχει και αυτή εργαστεί για το θέμα αλλά τώρα το θέμα είναι στα χέρια μας. Η δική μας Επιτροπή πρέπει να επαναπέμψει το θέμα στην Ολομέλεια. Και στο χρόνο που μας μένει λοιπόν μέχρι την ψηφοφορία πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δούμε τι ακριβώς μήνυμα θέλουμε να στείλει το Κοινοβούλιο προς τον έξω κόσμο. Είχαμε υποσχεθεί να καταλήξουμε σε μια πρόταση για τη μετανάστευση είδαμε ότι δεν, ήταν, δεν είχαν όλοι την ίδια δέσμευση και αντί να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας πρέπει να είμαστε πραγματικά επικοδομητικοί να καταλήξουμε σε συμφωνία και να έχουμε μια συνεπή μεταναστευτική πολιτική αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πράγματι διεθνής παράγων με κάποια αξιοπιστία και έξω από τα σύνορά της. Οι φιλελεύθεροι θα συνεργαστούν με την εισηγήτρια και ελπίζουμε στην δίμηνη αυτή διορία να μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτό το θέμα στην Ολομέλεια. Ε, Για να ξεκαθαρίσω τη διαδικασία, δεν θα ρίξω τώρα τη συζήτηση και θα καλέσω όλους να μιλήσουν, αλλά θα ζητήσω από τους συντονιστές των ομάδων να λάβουν το λόγο και η μόνη εξαίρεση είναι ο εισηγητής από την Επιτροπή Επασχόλησης και θα επανέλθουμε και στη δική μας εισηγήτρια. Διαφορετικά θα καταστερήσουμε πάρα πολύ από τους πρασίνους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ την κυρία Ματιά την εισηγήτρια. Πιστεύουμε ότι η πρότασή σας να ξεκινήσουμε με συνεδρίαση των σκιώδων ε, στη Λίμπε είναι κάτι πολύ καλό ως αρχή. Α ε, μην ξεχνάμε ότι προσπαθούμε εδώ να mm. καταλήξουμε, να έχουμε την πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να τονίσουμε ότι και εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να κατανοήσουμε αυτό το ζήτημα πριν αρχίσουμε το συμβιβασμό με του υπολείπου. Θέλουμε να διατηρήσουμε την συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης, αλλά βλέπουμε ε, ότι υπάρχει μια δυσκολία, γιατί για πρώτη φορά θα συναντηθεί στο τέλος αυτού του μήνα η Επιτροπή Απασχόλησης. Αν η πλειοψηφία εδώ λέει λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, τότε θα ήθελα να σας παροτρύνω να είστε σε πολύ στενή επαφή με τους συναδέλφους σας από τη δική σας ομάδα στην Επιτροπή Επασχόλησης. Εμείς θα προτιμούσαμε να έχουμε μία συνεργασία. Έχουμε ένα πρακτικό ερώτημα. Μετράμε αυτού του δύο μήνε από τώρα ή από πριν τα Χριστούγεννα. Φυσικά η προτίμησή μα θα είναι να μετράμε αυτό το χρόνο από σήμερα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μου είπαν ότι η κυρία Χάνη θέλει να μιλήσει εκ μέρου ομάδα τη. Ναι, εξ ονόντως Γκου έχω να σας πω τα εξή. Θέλουμε να εξετάσουμε το θέμα για άλλη μια φορά μαζί με την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, υπάρχουν πολύ σημαντικές ενδείξεις από την Επιτροπή Απασχόλησης που βέβαια έχουν αντίκτυπο και στη δική μας Επιτροπή. Δεν νομίζω λοιπόν ότι το θέμα είναι μόνο θέμα δικό μας και αυτό φαίνεται και από τον τίτλο και το περιεχόμενο της πρότασης. Δεν λοιπόν μόνο θέμα τη Επιτροπή Ελευθερών. Χρειαζόμαστε πολύ στην συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόληση. Και θα πρέπει να οργανωθούμε ανάλογα. Μια που προφανώ δεν υπάρχει προηγούμενο, μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε μεταξύ μα ποια θα είναι η άκουσα που θα ακολουθήσουμε. Εμεί προτείνουμε λοιπόν μαζί με την Επιτροπή περί ε, Απασχόληση να εργαστούμε και θα πρέπει βέβαια οι σκιώδει να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και για να είμαστε ειλικρινεί, θα ήταν καλό όλα τα θέματα που ήταν επιμαχόμενα καθ' όλη τη διάρκεια συζήτηση να ξανατεθούν επιτάπητο. Να δούμε από τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών της τελευταίας συνόδου πού υπήρχαν τα προβλήματα, τι θα πρέπει να είναι αντικείμενο νέων διαπραγματεύσεων και έτσι νομίζω θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε. Um, Ευχαριστώ. Γι' αυτό ποτέ δεν θα πιάσουν μια στην υπηρεσία πρωτοκόλλου γιατί μπερδεύω τη σειρά των ομάδων. Ο κύριος Κέρκο πρέπει να έχει πάρει το λόγο πριν. Ε, με συγχωρείτε. Ναι. Μην στεναχωριέστε όμως, γιατί και εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά. Αλλά η γενοδορή μου φτάνει τόσο μακριά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία <laughs> στην ΚΟΕΛ, όχι περαιτέρω, γιατί εγώ συμφωνώ με την προλαλή σας. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα που είναι θέμα της δικής μας Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και πάντοτε ε, είναι ενδιαφέρον όταν ε, άλλες ομάδες ασχολούνται και με το δικό μας έργο αλλά λυπούμε. Αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο και νομίζω ότι διαδικαστικά θα πρέπει να προέρχεται αυτό το έργο από τη ΛΥΜΠΕ και η ομάδα μου ανυπομονεί να προχωρήσει αυτό το ζήτημα το συντομότερο. Θα σας συνέβησαν στην Ολομέλεια ήταν ε, προφανή, ξέρουμε τι συνέβη. Τώρα είναι σημαντικό να ξαναπάμε όμω την έκθεση αυτή το συντομότερο στην Ολομέλεια για να προχωρήσει το ζήτημα, γιατί είναι σημαντικό. Και ο μόνο ε, τρόπο να το πράξουμε είναι να ασχοληθεί με το θέμα αυτό η Επιτροπή Λίμπε και να προσπαθήσουμε να μην αποκλίνουμε πάρα πολύ από αυτά που πιστεύουμε ότι ήταν σωστά να τεθούν στην Ολομέλεια. Σα ευχαριστώ, κύριε Σέρκα, από την Επιτροπή Επασχόληση, είναι ο Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ σήμερα γιατί έλαβα μια πρόσκληση από ένα πρόεδρο της Επιτροπής ΛΥΜΠ έτσι ώστε η Επιτροπή Επασχόλησης να μπορέσει να κάνει να ακουστούν και δικές της ε, σκέψεις ε, στα μέλη της ε, δικής σας Επιτροπής. Όπως είπε και κάποιος όλος ομιλήτης, εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Ένα θέμα διαδικασίας και ένα θέμα ουσιαστικό. Εγώ δεν θα μπω στο θέμα της διαδικασίας γιατί ε, υπάρχουν ε, οι αρμόδιοι που γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα και εγώ χάνομαι σε αυτές τις διαδικαστικές συζητήσει και επίσης ε, αποφεύγω αυτές τις εταιρικέ συζητήσεις μεταξύ των επιτροπών σαν την πανούκλα. Μένα με ενδιαφέρουν τα ουσιαστικά σημεία και τα ουσιαστικά σημεία είναι ότι αυτή η οδηγία έχει ένα τμήμα που αναφέρεται στα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης και εργασίας των επικών τρίτων χωρών που θα έρθουν να εργαστούν εδώ στην Ευρώπη και Εμάς μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε αν θα έχουν ίση μεταχείριση ή αν θα συνεχίσει να ισχύει η νομοθεσία της χώρας προελευσής τους. Αν δεν διευκρινιστεί σε αυτή την οδηγία η αρχή της, αρχής της ίσης μεταχείρισης, τότε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα σε ευρωπαϊκά επίπεδο για τα εργασιακά δικαιώματα γιατί ε, θα αποκλειστούν ορισμένοι ή ορισμένα δικαιώματα δεν θα εφαρμόζονται. Ε, υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα επί της ουσίας που θα το δούμε τα επόμενα χρόνια. Είδαμε τις δυσκολίες ε, που αντιμετωπίσαμε στο να δεκτεί κοινή γνώμη να κινηθούν στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης οι εργαζόμενοι βάσει της αρχής της χώρας προέλευσης. Τώρα έχουμε τον κινδύνου να υποβάλλονται στη νομοθεσία εξοκοινοτικών χωρών, αναπτυσσόμενων χωρών που ε, θα έρθουν να ε, φέρουν εδώ τη δική τους νομοθεσία. Αυτό είναι το ζήτημα, Πρόεδρε. Έτσι λοιπόν, ε, όποια λύση και αν δοθεί στη συνεργασία των δύο επιτροπών, αν είναι αρμόδια επιτροπή ΛΥΜΠΕ, ας λάβει υπόψη και αυτή την πολιτική διάσταση της οδηγίας και ας μην κοιτάξει αλλού, ας εξετάσει τα σοβαρά προβλήματα που έχει αυτή η οδηγία και εμείς είμαστε μικροί σε διάλογο. Ε, έστειλα και ένα email στην κυρία Ματιέ και τη το είπα. Είμαστε διατεθειμένοι λοιπόν να έχουμε ένα διάλογο γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για την οδηγία ως, ε, όπως μιλήσαμε για την οδηγία της ενέας άδεια, γιατί εδώ μιλάμε για την ίση μεταχείριση και πρέπει η αρχή αυτή να καταστεί πραγματικότητα, να μην μείνει στα λόγια. Ε, έτσι θα εργαστούμε τις επόμενες εβδομάδες, με οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε να εξεύρουμε επικοδομικές λύσεις που να ψηφιστούν και να εγκριθούν στην Ολομέλεια αλλά και να βοηθήσουν το ε, οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, στο μέλλον. Ε, γιατί δεν θέλουμε εδώ να τροφοδοτήσουμε την ξενοφοβία και τον ρατσισμό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωση. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ανεξάρτητα από την ε, απάντηση στην ερώτηση το πώς η εμπλοκή της Επιτροπής Απασχόλησης θα υλοποιηθεί, Τελικά η Ολομέλεια ψηφίζει. Έτσι λοιπόν όλα τα μέλη θα είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους. Σύμφωνα με το έγγραφό μου θα καλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια δήλωση. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει προσταμένη αξία. Εκτός και η Κομισιόν ε, έχει διακαή επιθυμία να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ματιέ για το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμή. και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο που μπορούμε επικοδομητικοί. Δεν έχω πολλά να πιστώσω εδώ, γιατί αυτά είναι θέματα που αφορούν τι αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου. Δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση επί σήμερα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ματιού. Δεν έχω τίποτα να απαντήσω κι εγώ συγκεκριμένο. Μόνο να σας πω ότι οπωσδήποτε θα είναι αποφεστική αυτή η εβδομάδα με τη συνάντηση μεταξύ των σχεδόν και μετά με τη συνάντηση με την Κομισιόν. Η κυρία Σεντίνη υπέβαλε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν ξέρω εσείς η γραμματεία έχει να απαντήσει. Από πότε ξεκινάει, ξεκινούν οι δύο μήνες κύριε Ματιό, φαντάζομαι από την ημέρα που ψηφίσαμε στην Ολομέλεια, στις 14 δηλαδή Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω. Okay, I'm, I'm, I'm told, I'm told, hang on, seen your request for floor. I'm told that it... Μου λένε ότι βασικά αρχίζει η διορία να τρέχει από τη στιγμή που αποφασίζει το Κοινοβούλιο, από τώρα δηλαδή. Όχι να σας πω κάτι, αφού αύριο συναντιούνται οι συντονιστές και φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες νομικές πτυχές που πρέπει να λυθούν, να περιμένουμε μέχρι αύριο, μέχρι να έχουμε όλες τις απαντήσεις. Άψογα. Συμφωνούν όλοι και όλες. Τελειώνει και το 5. Και περνάμε τώρα στο 6 ελάχιστες απαιτήσει για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη-μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα παρένθεση αναδιατύπωση. Η κυρία Γκυγιόμ. Σήμερα έχουμε την παρουσίασή της ε, για αυτό το αμφιλεγομενέστατο θέμα. Έχουν συναντηθεί πολλές φορές οι σκιώδεις μέχρι να συνταχθεί το κείμενο και όπως ξέρουμε uh, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δηλαδή θα υποβάλει αναθεωρημένη πρόταση τώρα και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η θέση προηγουμένως του Κοινοβουλίου. Και η διορία κατάθεσης τροπολογιών Λίγη στις 20 Ιανουαρίου το μεσημέρι. Πρώτα η εισηγήτρια και μετά η Κομισιόν. Ορίστε κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι, καλή χρονιά. Θα ήθελα καταρχήν να σας υπενθυμίσω μία διαπίστωση, ότι δηλαδή υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες ε, διαφορές μεταξύ των συστημάτων χορήγης ασύλου στην Ευρώπη. Το 2009 από 65% μέχρι 1% υπήρχαν τέτοιες διαφορές, ενώ οι διορίες για τη χορήγηση ή άρνηση έφταναν από τη μία μέχρι τις 30 μέρες. Οι διαφορές αυτές βέβαια υπάρχουν και ως προς τις ε, ε, λεγόμενες επιταχυμένες διαδικασίες. Τέτοιες ανισότητες βέβαια είναι ασυμβίβαστες με ένα, καθεστώς, με ένα κοινό καθεστώς ασύλου που πρέπει να έχει να έχει την ίδια ισχύ σε όλη την επικράτεια της Ένωσης εφόσον θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι ισότιμα και τα συστήματα μεμονωμένα που δεν είναι αλήθεια. Άρα μόνο η εναρμόνιση των συστημάτων και οι εγγυήσει τους μπορούν να καταλήξουν σε ένα κοινό σύστημα. Μία δεν νομοθετική τέτοια εναρμόνιση είναι απαραίτητη γιατί μία απλή συνεργασία όπως θεωρούν ορισμένοι δεν αρκεί. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσουμε σε βάθος την οδηγία ώστε να μπορέσει επιτέλους να υπάρξει μία προσβατή και δίκαια και αποτελεσματική οδηγία. Υπάρχουν πολλές ιδέες, το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε το γνωρίζω κι εγώ. Ιδιαίτερα, για να το πω ρητά, το κόστος των διαδικασιών αυτών είναι ο λόγος των διαφωνιών. Πράγματι υπάρχει κόστος, αλλά παρακαλώ τους συναδέλφους και τους προσώπους του Συμβουλίου να σκεφτούν και κάτι άλλο που για μένα αποτελεί πεποίθηση ότι η κακή χρήση των διαδικασιών είναι εκείνη που αυξάνει το κόστος για τα κράτη-μέλη. Αυτό το δείχνουν και οι καθυστερήσεις της διαδικασίας προσφυγής μεταξύ άλλων. Πρέπει λοιπόν να διευκολυνθούν και να βελτιωθούν οι διαδικασίες αυτές για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα γιατί αυτή τη στιγμή βλάπτονται όχι μόνο τα κράτη-μέλη αλλά και τα θύματα. Μία ποιοτική απόφαση θα έπρεπε να επιτρέπει την λήψη υπόψη όλη τη πραγματικότητα που αφορά τον ετούντα και να ε, ακολουθείται από πλήρη δικαιολόγηση της έγκρισης ή απόρριψης του αιτήματο, να υπάρχει καλύτερη ταύτιση των προβλημάτων και να υπάρξει και μειωμένο κόστος για τα κράτη-μέλη εφόσον μάλιστα ιδιαίτερα στην περίπτωση που θα χρειαστεί να επαναπέμψουν τον ετούντα στο κράτος προέλευσής του. στην ουσία πρόκειται για τη βελτίωση ορισμένων συγκεκριμένων πτυχών της διαδικασίας όπως μεγαλύτερη συνοχή ως προς το ποια είναι κάθε φορά η αρμόδια αρχή και ποια είναι η τελική αρχή που καθορίζει τη λήψη της απόφασης και έπειτα ποιες είναι οι ελάχιστες προβλεπόμενες διαδικασίες όπως προβλέπει και, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα πληροφόρηση, το δικαίωμα να ακουστεί κανείς στο δικαστήριο, η νομική βοήθεια και αρρωγή και έπειτα να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των ετούντων, ιδίως δε των παιδιών τους ή να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα εργαλεία που ήδη διαθέτουμε όπως οι τρίτες χώρες σουρ και τέτοια. Έτσι τελειώνει μία πρώτη φάση συνεργασίας με τους κοιόδης τους οποίους ευχαριστώ συλλήβδιν για τη συνεργασία τους και νομίζω και ελπίζω ότι αυτά θα βοηθήσουν όλους και όλες για να αντιμετωπίσουμε και να συγκρίνουμε τις αντιμετωπίσεις που έχουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους για να δούμε ποιες είναι οι διαφορές γιατί το θέμα είναι σημαντικό ιδίω ω προς τον ανθρώπινο του χαρακτήρα. Από την Επιτροπή και μετά την Ολομέλεια θα σας, δι... θα σας ε, δώσω υποδείξεις και θα προσέχω πάντοτε ιδιαίτερα όπως το κάνω πάντοτε για να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Δύο άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Βλέπω και πολλοί άλλοι. Προστίθενται. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Βέξτρου. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την συγχύτρια για όλες τις προσπαθίες της. Ε, εγώ δεν είμαι σκιώδης ε, γι' αυτό το φακέλο, αλλά καθώς ε, είμαι συγχύτρια για την αναδιατύπωση του Δουπλίνου 2, Προσπαθώ να συσχετίσω όλους αυτούς τους φακέλους. Καλωσορίζω την πρόταση της Κομισιόν, όπως και την εκθέση της κυρίας Γιώμ έθεσε, παρουσίασε πάρα πολλέ φιλόδοξε τροπολογίε. Ε, θέλω να επιστήσω την προσοχή σα ότι την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο μία προφορική ερώτηση για το κόστο ε, τη εξέταση των ε, αιτήσεων ασύλου στα κράτη-μέλη θα συζητηθεί. υπομονώ να δω την απάντηση του Συμβουλίου γιατί υπάρχει μεγάλη απόκληση μεταξύ των διαδικασιών των κρατών μελών και έχουμε πολλά διαφορετικά αποτελέσματα για τους ετούντες άσυλο και υπάρχουν πάρα πολλέ επιφυλάξει ε, για το φάκελο αυτό στο Συμβούλιο. Και επομένω θεωρώ ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε εμεί στο Κοινοβούλιο το σημαντικό μα έργο και να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Άλλωστε έχουμε μία κοινή πρόθεση να αντιμετωπίσουμε μέχρι το 2012 και θέλω να ευχαριστήσω και την κυρία Γκυγιόμ για όλα όσα έκανε με αυτό το ζωτικό ζήτημα. Ευχαριστώ κύριε Φίξτρομ. Κύριε Φλότρα, και κατόπιν ο κ. Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω ενθερμα την κυρία Κιγιόμ. Νομίζω ότι είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε μια η συγγετρία η οποία συνειδητοποιεί τις δυσκολίες που απομένουν για να έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που να παρέχει αποτελεσματική προστασία. Η έκθεσή της ε, υποστηρίζει τις προτάσεις αναδιατύπωσης της Κομισιόν και μάλιστα εμβαθύνει και σε κάποιες προτάσεις και τις αναπτύσσει κυρίως ό,τι αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά ε, τις ε, αρμόδιες αρχές. Επίσης, ε, για το να έχουμε έναν ορισμό για τα μέλη της οικογένειας, ε, για το να έχουμε συστηματική ενημέρωση ε, σε μία γλώσσα που να καταλαβαίνει ο ετών ε, επίσης ε, έχουμε και άλλα σημεία πολύ σημαντικά όπως είναι το να έχουμε την κατάργηση της ασφαλούς τρίτης χώρας, το να υπάρχει προθεσμία για την προσφυγή. Νομίζω ότι όλα αυτά τα στοιχεία που συνεισφέρει η πρόταση κυρίας Γιώμη είναι εξαιρετικά και τα υποστηρίζουμε πιθανότητα για ορισμένα σημεία θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Αναφέρομαι στην ικανότητα των μη κυβερνητικών οργανώσεων από την αρχή να έχουν πρόσβαση και όχι αναλόγω με τη βούληση των κρατών μελών για να μπορούν να ε, συνοδεύουν και να παρακολουθούν τη διαδικασία ε, της αίτησης από την αρχή επίσης ε, δεν θα πρέπει τη διαδικασία να, την, να βαρύνει τον Τούτα επίσης ε, θα πρέπει να έχουμε και τις ε, ε, ιατρικές εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και να ερμηνεύονται προς όφελος του ετούντα. Το Συμβούλιο φαίνεται να έχει μία θέση μη υπεύθυνη και εγώ νομίζω ότι η δουλειά του Κοινοβουλίου θα αναγκάσει το Συμβούλιο να αποκαλύψει αυτά τα κακά επιχειρήματα επιχειρήματα που αφορούν και το κόστος, ε, γιατί ε, κοστίζει το να κλείνουμε στα κέντρα κράτησης ε, τους ετούτες και επίσης έχουμε και μια διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων που κοστίζει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, αν πείσουμε το Συμβούλιο για αυτή τη διαδικασία θα ωφεληθούμε τα μάλα. Ευχαριστώ κύριο Τριανταφυλίδης και κατόπιν κύριε Χολμαϊρ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την κυρία Γκυγιόμ για την εξαιρετική της έκθεση, κυρίως ε, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που διακυβεύονται θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, πολύ επικοδομητική στάση που είχε γιατί συζητήσαμε με τους σκιώδες συζητητές ε, τις προτάσεις άρθρο προς άρθρο και συναντήθηκε και με τον καθένα μεμονωμένα. Υποστηρίζω τις προτάσεις καθώς συμφωνώ με τη διάκριση της μεταξύ της ε, αρμόδιας αρχής και της determining authority. Επίσης νομίζω ότι η νομική ερωγή θα πρέπει να προβαίνει και στην προετοιμασία των διαδικαστικών εγγράφων και το βάρος της απόδειξης πρέπει να το έχει η αρχή που λαμβάνει την απόφαση και όχι η αρχή στην οποία απευθύνεται η αίτηση. Επίσης, ε, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην διαγραφή του άρθρου που έχει να κάνει με τις ασφαλείς χώρες. Και επίσης, ε, για την πρώτη χώρα, η χώρα πρώτης κατάθεσης ασύλου θα πρέπει να καθορίζεται και ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίσταση στην οποία βρίσκεται το ετών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και που ήσασταν και στην κυρία Χολμάιερ και μετά κυρία Χίρς. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια για την υποβολή αυτή τη έκθεση και για τις πολλές συνομιλίες που είχαμε με την εισηγήτρια. Πολύ αντικειμενικά. Το θέμα της ασυλίας και της μετανάστευσης είναι κάτι που δεν θα μας απασχολήσει μόνο όσον αφορά τι διάφορε επιμέρου οδηγίε, αλλά και όσον αφορά την φτώχεια και την κατάσταση σε πολλέ χώρε του κόσμου. Πού θα μα θέλουν συνεχώ ενώπιον νέων προκλήσεων. Θα ήθελα ιδιαίτερα να χαιρετήσω στην έκθεση της κυρίας Γκυγιόμ το ότι τονίζει ιδιαίτερα το θέμα των παντρεμένων ανηλίκων και ένα θέμα που συζήτησα και με την κυρία Ζεν Τζιν Λάμπετ δεν επιτρέπεται δηλαδή παιδιά που έχουν εξαναγκαστεί να παντρευτούν να μην έχουν πρόσβαση σε ε, νομική εκπροσώπηση. Κάθε ε, άτομο θα πρέπει να έχει έναν νομικό εκπρόσωπο που θα προασπίζει τα δικαιώματά του. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό. Έχω βέβαια και κάποιε επιφυλάξει και το ξέρει η κυρία Γεγιόμ πάνω στην πρόταση τη Κομισιόν. Καταρχήν μου φαίνεται πολύ αφίβολο ότι οι νεπαρκεί διαδικασίε είναι εκείνε που οδηγούν σε υψηλό κόστο. Γιατί αν δούμε παραδείγματο χάρη τι γίνεται στην Ελλάδα, το υψηλό κόστος δεν προέρχεται από κακές διαδικασίες, από τον τεράστιο αριθμό ζητούν άσυλο που έχουν έρθει εν μέρη και παράνομα στη χώρα αυτή. Και πολλοί από αυτούς ε, ε, δεν θέλουν καν ασύλο, αλλά έρχονται ανοιχτά και ελεύθερα όπως φαίνεται στην Ελλάδα για διάφορους άλλους ανθρώπινους λόγους λόγω ε, ένδυας λόγω του ότι ελπίζουν να έχουν μια καλύτερη μια καλύτερη ζωή. Κοιτάξτε, με, με, η πρόταση λέει παρακαλώ συντομεύεται. Κοιτάξτε, είναι η πρώτη ζήτηση που έχουμε το θέματος. Ναι, ναι, προσπαθώ, προσπαθώ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω σε δύο λεπτά όμως. Έχουμε χρόνο, γιατί βιαζόμαστε. Α, προσπαθώ να είμαι δίκαιο όμως για όλους. Άμα δεν θέλετε, Όχι, δεν ολοκληρώνω εδώ. Δεν, δεν τελειώνω εδώ. Θα σα πω αυτά που έχω να πω. Δεν μου φαίνεται ότι είναι δίκαιο να μου πείτε να κλείσω εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω. Όσον αφορά το θέμα του νομικού εκπροσώπου χωρίς κόστος έχω επιφυλάξεις ε, έχω επίσης επιφυλάξεις το ότι αιτήσει οι οποίες δεν αιτιολογούνται σωστά δεν μπορούν να επιταχυνθούν όπως το παρελθόν. Επίσης έχω κάποιες επιφυλάξεις για τον ορισμό του ετούντος που δεν πρέπει να είναι με να είναι στην, να είναι συγγνώμη πίκος εν λόγω χώρας. Υπάρχει όμως το πρωτόκολλο Ασνάρ ότι όταν κάποιος ε, πάει σε μια άλλη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητήσει εκεί άσυλο. Αυτό δεν είναι δυνατό γιατί θεωρούμε ότι και 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τηρούν και σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Μετά, το ορισμός των μελών της οικογένειας. και θέματα ε, όσον αφορά την απόρριψη μιας αίτησης, την εξέταση της άρνησης για ιατρική εξέταση και επίσης την στροφή του δικαιώματος του βάρους απόδειξης ότι μετά από έξι μήνες θα πρέπει το κράτος να αποδείξει κατά πόσον ένας ετών άσυλο έχει πραγματικά ανάγκη ή όχι. Αυτό μου φαίνεται πολύ ε, προβληματικό. Λοιπόν, έχουμε νομίζω ανάγκη να συζητήσουμε εις, βάθος το θέμα και σε ευχαριστώ που ακούσατε. Πρόεδρος, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα και ότι πρώτη, είναι η πρώτη συζήτηση αυτή. Αλλά αν συμφωνήσουμε να έχουμε περιορισμένο χρόνο ε, αγόρευσης, όλοι έχουν δύο λεπτά και εσείς έχετε πέντε, όλοι θα θέλουν το ίδιο. Η κυρία Χίρς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έγινε μια καλή αρχή νομίζω με την έκθεση αυτή. Χαίρομαι που την έχουμε στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία. Οπωσδήποτε υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν. Είναι σαφές, θα το επιδιώξουμε αυτό και με τροπολογίες. Αλλά μου φαίνεται είναι πολύ καλό και σημαντικό μήνυμα ότι θα πρέπει όλη τη δέσμη για το άσυλο να την περάσουμε λίγο πολύ ταυτόχρονα γιατί καταρχήν θα πρέπει να έχουμε τους ίδιους ορισμούς και στις όλες τις οδηγίες, να μην έχουμε απόκληση των ορισμών. Εκτός αυτού να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το Συμβούλιο, να πούμε ότι θέλουμε και αυτή την οδηγία για τη διαδικασία. Γιατί θεωρώ ότι όταν έχουμε μία γλίγορη και καλή διαδικασία και δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο αποκλείουν το μεν όταν το έχουμε αυτό θα βοηθήσουμε και τις δύο πλευρές και την χώρα υποδοχής γιατί σύνομα θα υπάρχει διευκρίνηση αλλά και για τον ετούντα άσυλο. Δεν θα είναι δηλαδή τρία-τέσσερα χρόνια σε μια χώρα, θα έχει εγκατασταθεί καλά εκεί, θα έχει ε, ξεκινήσει να δημιουργεί τη ζωή του και μετά θα το πούμε όχι, θα πρέπει να πας πίσω από εκεί όρθες. Λοιπόν, βραχυπρόθεσμα ίσως θα είναι υψηλότερο το κόστος για τα κράτη-μέλη, αλλά μακροπρόθεσμα μια καλή διαδικασία θα αξίζει πραγματικά. Ακόμα και αν εξτάσουμε το θέμα από την ε, οικονομική πλευρά, ένα θέμα που τίθεται από τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο συνεχώς. Λοιπόν, εάν αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να έχουμε δυνατότητα ασύλου, θα πρέπει να είμαστε και δίκαιοι και να μην προσπαθούμε να ανοίξουμε ε, κάποια παραθυράκια ούτως ώστε να παρεμποδίσουμε τα άτομα αυτά που έχουν ανάγκη να έρθουν στις χώρες μας. Λοιπόν, αν πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ του ασύλου θα πρέπει να έχουμε την τόλμη να υιοθετήσουμε οδηγίες και να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε συνεπείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χίρσλε Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο η κυρία Γκέ, αν το προφέρω σωστά το όνομά σας, και ο κύριος Κούντς έχουν ε, εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκυγιόμ για το σχέδιο έκθεσης. Νομίζω ότι συνόψεις ε, πολύ καλά τα κυρία στοιχεία και το γενικό πνεύμα της πρότασης της, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήδη είχαμε την ευκαιρία του φθινόπωρο να επανέλθουμε ε, στις εξηγήσει της πρότασης. Επίσης, κάνουμε και μια αξιολόγηση της σημερινής οδηγίας που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο και που υποστηρίζει επίσης το σκεπτικό μας. Προκειμένου να έχουμε μια ταχύ διαδικασία και αποτελεσματική διαδικασία αλλά και εξασφάλιση της ποιότητας. Και χαίρομαι που οι προλερίσοντες ε, ανέφεραν ε, ότι η ιδέα του front-loading ε, είναι κάτι αποδοτικό, κάτι που μας ωφελεί και για το θέμα του κόστους θα επανέλθουμε στην Ολομέλεια βάσει και της προφορικής ερώτησης που λάβαμε. Όπως είπατε, έχουμε δεσμευτεί να βάλουμε μια αναθεωρημένη πρόταση βάσει των σημαντικών δυσκολιών που απαντήθηκαν πριν την έναρξη της Πολωνικής Προεδρίας. Οι δυσκολίες ε, στο Συμβούλιο είναι υπαρκτές και για αυτό το λόγο είναι όλο ένα και πιο σημαντικό να έχουμε και την ε, γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου που επί του φακέλου αυτού θεωρώ ότι θα μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο για να επηρεάσει την πρότασή μας. Πέραν αυτών, η αλήθεια είναι ότι σημειώσαμε ότι το σχέδιο έκθεση της κυρίας Γκυγιόμ ε, υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση της Κομισιόν. Σε ορισμένες ε, πτυχές ε, δεν σας κρύβω ότι και εμείς ως Κομισιόν είχαμε κάποια προβλήματα χωρίς καν να αφαιρθούμε στο πρωτόκολλο ΣΝΑΡ, για μας είναι προφανές ότι πρέπει η οδηγία να ισχύει και για τους, οπικό, για τους οπικούς των τρίτων χωρών ε, υπόψη της νομικής βάσης ε, του άρθρου 58 της συνθήκης. Ορισμένες ε, τροπολογίες θέλουν να ενισχύσουν τις δικονομικές εγγύησεις, ίσως πέραν ε, του πνεύματος της Ευρωπαϊκής Νομολογίας, ε, του Δικαστηρίου του Στρασβούργου και του Δικαστηρίου του Ξεμβούργου, αλλά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε αυτά τα, στοιχεία περαιτέρω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επανερχόμαστε στην κυρία Κιγιό. Ναι, σας ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Έχουμε και χρόνο, τέλεια. Όπως ε, υπόθηκε μόλις, γνωρίζουμε ότι η μέσα σε έξι μήνες ε, η Κομισιόν θα παρουσιάσει θεωρημένες ε, να παρουσιαστούν προτάσεις ε, για την οδηγία αυτή κατά αλλά και για τη διαδικασία. Για τη διαδικασία. Θέλουμε να πλουστεύσουμε μία διατύπωση που μας φάνηκε ιδιαίτερα πολύπλοκη και να αποφύγουμε να μπλοκαριστούν συζητήσεις στο Συμβούλιο. Εγώ συμφωνώ με πολλά πως ακούστηκαν εδώ. Πίστευω ότι μου σαφείς προηγούμενος, θα το ξαναπώ όμως. Δεν πρέπει εδώ ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφύγει να αναλάβει τις ευθύνες του. Το αντίθετο, θα πρέπει να λειτουργήσει ο συνομοθέτης πλήρως αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα φιλοδοξίας, δεν πρέπει να παρατηθούμε. Πιστεύω ότι το επίπεδο προστασίας ε, για όσους το χρειάζονται αλλά και οι δικονομικές και οικονομικές δυσκολίες ε, που ε, και βεβαιότητες από το τα κράτη-μέλη πρέπει να τεθούν στο στόχαστρο. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος για το 2011 για να σεβαστούμε τις προθεσμίες. Δεν θα έπρεπε να καταλήξουμε σε ένα αποδυναμωμένο κείμενο ή ένα κακές ποιότητας κείμενο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υιοθετήσει μια ζωτική θέση για να δοθεί συνέχεια σε αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ για την έκθεση αυτή. Να επιθυμίσω στους συναδέλφους ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 20 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Περνάμε στο σημείο 7 της αλλά και τι απαιτήσει για την αναγνώριση και το καθεστώ των επικών των ε, τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ω δικαιούχων διεθνού προστασία και το περιεχόμενο της περιεχόμενης προστασία. Με διατύπωση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Λάμπερτ που οργάνωσε μια δεύτερη συνεδρίαση με τους Κιώδες για να συζητηθούν πιθανή συμβίβασμα για τις τροπολογίες στην έκθεσή της και για να προετοιμαστούμε για την ψηφοφορία προσανατολισμού που έχει τεθεί περί τα τέλη Ιανουαρίου. Κυρία Λάμπερτ, παρακαλώ μπορείτε να πάρετε το λόγο να μας αναφέρετε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις συζητητές για τη συνάντηση που είχαμε το Δεκέμβριο Πιστεύω ότι τότε είδαμε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί που αφορούν και το τομέα και το περιεχόμενο της προστασίας. Θα θυμάστε ότι η οδηγία αυτή έχει να κάνει με δύο τεινά. Το θέμα της αναγνώρισης που αφορά την διαδικασία και προστασίας και έχουμε και το τμήμα του περιεχομένου και τι δουλειά πρέπει να κάνουν το κρατημένο για την παροχή αυτής της προστασίας. Δύο τμήματα λοιπόν και το κύριο ζήτημα είναι ότι η διατύπωση προσπάθησε να ε, συμφωνήσει αυτά τα δύο καθεστώτα υπό το άρθρο 9 και μιλάμε για το καθεστώς ε, των προσφύγων και στο άρθρο 15 μιλάμε για την επικουρική προστασία όπως την έχουμε αυτή τη στιγμή όσους δηλαδή βρίσκονται σε κίνδυνο βλάβης. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, σε ποιο βαθμό πρέπει να έχουμε διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων αυτών. Είχαμε μία πολύ σύντομη συζήτηση όταν κατατέθηκαν οι τροπολογίες, τότε είπα ότι τι ήθελα εγώ να κάνω με τις τροπολογίες. Ήθελα να αναφερθώ στα σημεία που είχαμε και στην αναδιατύπωση και θέλαμε να αναφερθούμε και όσοι όσα δεν αναπτύσσαν στο πεδίο εφαρμογή της αναδιατύπωσης. Και πρέπει να δούμε αν ε, για όσα είναι εκτός υπάρχει ουσιαστική πολιτική συμφωνία με αυτή την Επιτροπή. Είναι χρήσιμη λοιπόν η σημερινή συζήτηση ως προς αυτή την κατεύθυνση. Και θα αναφερθώ σε αυτά τα σημεία σε λίγο. Στη σημεία που φαίνεται να μπορούμε να βρούμε τώρα μια συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων ως προς τα δικαιώματα έχει να κάνει με το άρθρο 23, δηλαδή για τις ευπαθείς ομάδες, τις οβάλλοντες ομάδες και εδώ 769 συμβιβασμό θα έχουμε πιθανότατα σε σχέση με το τι θα κάνουμε για το βέλτιστο συμφερόν του παιδιού. Άρθρο 25 και τα σχετικά εκτιμώντα. Επίσης είχαμε χρήσιμη συζήτηση για το θέμα των μέτρων ένταξης, ε, άρθρο 34, εκτιμώντα 39 και Βλέπουμε και τις ε, τροπολογίες ε, ότι είναι καθήκον των κρατών μελών ε, να προβούν σε αυτή την προσφορά. Δεν πρέπει να είναι απέτηση εδώ, αλλά Αν υπάρχουν ε, και ευτερίες παροχές ανθρωπιστικής προστασίας, ε, θέλουμε να τις ε, αδράξουμε αυτές τις δυνατότητες, γιατί εμείς πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο πόσο σημαντικά είναι τα θέματα, τα μέτρα για την ένταξη. Επίσης, έχουμε κάποια συμφωνία για θέματα σχετικά με το φύλλο. Εκεί έχουμε αρκετές τροπολογίες, 26-27 έχουν να κάνουν και με τα σχετικά εκτιμώντας και με το διατακτικό. Τώρα, το τομείς συζήτηση όπου δεν είχαμε ακόμη την ευκαιρία να εξετάσουμε λεπτομερώς τις ε, συναντήσεις των σκιώδων είναι σχετικά με θέματα που αναφέρθηκαν σε άλλα μέτρα. Έχουμε τα θέματα που αφορούν τον ορισμό της οικογένειας. Αυτό δεν το συζητήσαμε ως και ακόμα. Και υπάρχουν αρκετές ε, τροπολογίες ε, από την 39 ως τη 43 που έχουν να κάνουν με το θέμα των έγαμων ενηλίκων κτλ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η οδηγία δεν έχει να κάνει με οικογενειακή επανένωση εδώ μιλάμε για μέλη της οικογένειας και αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι παρόντες στην επικράτεια τη στιγμή που ζήτησαν ε, άσυλο ή άλλες μορφές ε, ανθρωπιστικής προστασίας. Δεν μιλάμε για επανένωση λοιπόν. Υπάρχουν και αποκλήσει απόψει εδώ. Έτσι λοιπόν, εγώ θέλω να σα πω ότι θέλω να διατηρήσω πιο ευρύ τον ορισμό αυτό. Υπάρχουν ε, κάποιε περιπτώσει που σχετίζονται με το θέμα των αγαπημένων υλίκων. Έχουμε πολύ μικρέ τέτοιε, πολύ μικρό αριθμό τέτοιων περιπτώσεων, αλλά αν δεν το ρυθμίσουμε αυτό θα αφήσουμε σε ένα νομικό κενό του ανθρώπους αυτούς. Γιατί μάλλον θα του αντιμετωπίσουν όχι ως ανήλικους, αλλά ως παντρεμένους. Και μπορεί αυτό να προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες αλλά φυσικά ενδιαφέρομαι να ακούσω και τι απόψει τη επιτροπή από αυτού. Έχουμε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με το άρθρο 7, Τροπολογίε 46 46-52 και εδώ υπάρχει απόκληση απόψεων. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με το εξή, αλλά δεν υπάρχει στην διατύπωση το αν ε, μόνο ένα κράτος μπορεί να προσφέρει την προστασία, αλλά η οδηγία επιτρέπει και στις διεθνείς, στους διεθνείς οργανισμούς. Και βλέπουμε ότι πώς μπορούν άλλοι φορείς ε, να θεωρηθούν ως αποτελεσματική παροχής ε, προστασίας, πάροχη προστασίας. Επίσης, έχουμε τροπολογία για το θέμα της προστασίας και μπορούμε να βρούμε ένα συμβασμό για τις τροπολογίες 53 και 54. Επίσης, θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας για το άρθρο 5.3, τροπολογία 44-45, λεμπρινίδης κτλ. Για τις περιστάσεις βάσει των οποίων πιστεύτηκε ότι οι άνθρωποι έδρασαν ε, με έναν τρόπο ε, για να, κάνουν, ε, να, να, γίνει πιστευτό ότι χρειάζεται προστασία όταν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και το θέμα του πεδίου εφαρμογή συνολικά για το αν έχουμε εδώ ε, τους υπηκόους μονοτρίτων χωρών ή ανασχολούμαστε με όλες τις περιπτώσεις. Τροπολογία 34 της κυρία Γιώργη Νομίζω ότι θα, ήταν ε, πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τις απόψεις διαφορών μελών. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες, 106. Δεν θέλω τώρα εδώ να εξαντλήσω την υπομονή σας, αλλά αν φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, είτε μπορούμε να τις δούμε εδώ, είτε εκτός. Ευχαρίστως να το συζητήσουμε κι αλλού. Thank you very much. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Έχουν ζητήσει δύο το λόγο. Θέλει κανείς άλλος ή καμία άλλη. Καλά, τρεις τώρα, τρεις. Η κυρία Βίκ Στρόμ. Ευχαριστώ πολύ και την ησυχήτρια για όλα όσα έκανε για αυτό το θέμα καθώς και για την συμπερίληψη όλων των πτυχών που έλαβε υπόψη στο κείμενό της. Δέχομαι την πρόταση της Κομισιόν και την έκθεση αυτή και πρέπει να συνεχίσουμε να προχωρούμε με το θέμα όπως και κατά υπόλοιπα εξάλλου. Ας τονίσω όμως μερικές από τις τροπολογίες που δεν δέχτηκε, δεν συμπεριέλαβε η εισηγήτρια. Μαζί με συναδέλφους είχα καταθέσει τροπολογίες για τα δικαιώματα των παιδών με βάση τη σύμβαση του ΟΗΕ για αυτό το θέμα και είχα ζητήσει επίσης να υπάρξει γλωσσική εκπαίδευση για να διευκολύνει αυτό την ε, συμμετοχή των μεταναστών στις χώρες όπου ζουν καθώς και αναφέρθηκα στα θέματα των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που έχει ο καθένας. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω αυτήν την τροπολογιούλα που νομίζω όμως ότι μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λαμπέρ. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η οδηγία μαζί με την προηγουμένη αποτελούν μια δέσμη μέτρων για τους οποίους δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ομάδων. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ των ε, θέσεων που πρέπει να γεφυρωθεί και είναι δύσκολο να φτάσουμε στη συμφωνία γιατί είναι φιλόδοξη οδηγία. Η πρόταση της Κομισιόν είναι φιλόδοξη. Γιατί? Για να διατύπωση, για να διάφραση το περιεχομένο της Διεθνού προστασίας σε συνδυασμό με το καθεστώς ε, του πρόσφυγα είναι κάτι φιλόδοξο. Πέρα από τις τροπολογίες ε, που θα μπορούσαν να είναι ίσον ε, ω σημασία κατά την άποψή μου, εδώ νομίζω ότι το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στη συμφωνία. Και το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Τι συμβαίνει με τους πρόσφυγες. Πώς ε, ερμηνεύει τον όρο πρόσφυγα στη Σύμβαση της Γενέβης. Είναι πολύ αυστηρή η ερμηνεία. Γιατί, κοιτάξτε, εγώ πρέπει να αναφερθώ στον καταβλισμό της Χαφάρ που επισκέφτηκα εγώ γιατί επισκέφτηκα αυτούς τους καταβλισμούς που υπάρχουν στη Μάλτα, τους τρεις, ε, ε, ένα από τον καταβλισμό υπήρχε μόνο ε, μία οικογένεια και μία γυναίκα από τη Λιβύη και από άλλη χώρα που είχαν το καθεστώς του πρόσφυγα και οι υπόλοιποι προέρχονταν από τη Σομαλία και είναι φυγάδες από τη Σομαλία. Δηλαδή είναι, δεν είναι άτομα που δεν να κρατηθούν ε, όταν φτάσουν. Δεν είναι πολιτικοί πρόσφυγες, αλλά απλώς ε, προσπαθούν να αποφύγουν την απειλή του πολέμου και άλλοι έρχονταν ε, από το Σουδάν ε, το άλλο 50%. Ε, έτσι λοιπόν, αν βλέπουμε το ζήτημα έτσι, νομίζω ότι δεν βλέπουμε συνολικά το πρόβλημα. Η ε, ίδια η Επιτροπή που είναι αρμόδια για τους πρόσφυγες, η Πατερμοστία για τους πρόσφυγες, μπορεί να μας επιβεβαιώσει αυτά τα δεδομένα για τους μετανάστες στη Μάλτα. Γιατί, κοιτάξτε, εμείς το πρόβλημα που έχουμε στην Ευρώπη είναι πρόβλημα συνόρων. Και είχαμε εδώ και τον κύριο Κοτερίος που μίλησε για τους ε, ε, πρόσφυγες στον κόσμο, αλλά τώρα εδώ εμείς συζητούμε πώς εμείς ε, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των Ετήσιο ασύλου. Ένας ε, ετών ε, πρέπει να δώσει τα δακτυλικά του αποτυπώματα και όταν ε, προσπαθεί να φτάσει στον προορισμό που ονειρεύεται που είναι η Σουηδία δίνει τα δακτυλικά του αποτυπώματα στη Μάλτα και έχουμε κάποιους που ήδη έχουν επιστραφεί τρεις και τέσσερις φορές. Έτσι λοιπόν ε, δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την ε, κατάσταση με τους οικονομικούς μετανάστες που παίρνουν ε, ένα εισιτήριο στην, στο Εκουαδόρ ή σε άλλη χώρα και δεν βρίσκονται στην ίδια θέση. Πρέπει να το δούμε αυτό, δηλαδή είναι ουσιαστικό το θέμα. Πρέπει να δούμε την κάθε συγκεκριμένη περίσταση και αυτό το πρόβλημα τι ουσιαστικά κάνουμε με αυτού του 1500 που υπάρχουν τώρα στη Μάλτα, παραδείγματο χάρη, άλλου τόσου μπορεί να είναι στην Ελλάδα. Ούτε καν ε, τα στοιχεία δεν έχουμε. Και τι μπορούν να κάνουν τα 27 κράτη-μέλη, πώ μπορούν να έχουν μια αλληλέγγυα πολιτική για το θέμα αυτό. Okay, thank you. Next on my list, Mrs. Ευχαριστώ κύριε Χολμαϊέρ. Δεν θέλω να σας τρομοκρατήσω άλλη μια φορά κύριε Πρόεδρε μακρηγορώντας αλλά θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Τζιν Λέμπε για τις πάρα πολλές και πολύ επικοδομικές συνομιλίες που είχε μαζί μας. Προσπαθήσαμε να αναφερθούμε σε ορισμένα θέματα όσον αφορά το περιεχόμενό του Μια από αυτή που δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε μέχρι το τέλος είναι το θέμα της χορήγησης της ε, προστασία υγείας. Λέγεται ότι θα πρέπει η προστασία της υγείας αυτή να γίνεται όπως δίνεται και στους άλλους πολίτες της χώρας αυτής. Αλλά βέβαια υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο τι δικαιώματα έχει στον τομέα αυτό ένας πολίτης ε, στα διάφορα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Εγώ θα ήθελα να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα, ελάχιστη χορήγηση ή ιατροφαρμακευτικής προστασίας Ακριβώς γιατί τα συστήματα διαφέρουν τόσο πολύ από χώρα σε χώρα που δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική διατύπωση. Γιατί σε ορισμένε χώρε υπάρχουν 100% ιατρική προστασία μέχρι μεταμόσχευση. Σε άλλες χώρες ε, δεν αναγνωρίζεται καν μια γενική θεραπεία σε ένα νοσοκομείο. Παραδόν χάρη υπάρχουν χώρε όπω η Ισπανία, η Γερμανία, η Αυστρία που αναγνωρίζουν πολλά, άλλε χώρε τίποτα σχεδόν. Λοιπόν θα πρέπει να αναφέρουμε σε ένα ελάχιστο ένα ελάχιστο πρότυπο που θα πρέπει να ε, ε, τηρείται για να δείξουμε έτσι το σεβασμό μας προς τους αιτούντους ε, αυτούς άσυλο. Συμφωνώ με την κυρία Τζιν Λάμεθ όσον αφορά τον ορισμό της οικογένειας. Υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της οικογένειας στις διάφορες οδηγίες και αυτό είναι προβληματικό. Δεν μπορεί σε κάθε οδηγία να έχουμε άλλο ορισμό της οικογένειας. γιατί οι αρχέ μετά δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν αυτά. Χρειάζονται έναν σαφή ορισμό της οικογένειας παντού τον ίδιο. Και ε, συμφωνώ ότι αυτή η οδηγία δεν ασχολείται με την επανένωση των ε, οικογενειών, αλλά με τον ορισμό των ελαχιστών προτύπων για την αναγνώριση. Όχι μια οδηγία που ασχολείται γενικά με την επανένωση των οικογενειών. Υπάρχει βέβαια και ένα πρόβλημα όσον αφορά τον διαχωρισμό των συμπληρωματικών δικαιωμάτων και εκείνων που προβλέπονται ε, σαν προστατεύσιμα δικαιώματα από την ε, συνθήκη της Γενέβης. Αυτό θέμα οπωσδήποτε θα μας απασχολήσει ήδη μακρόν ακόμα και πάρα πολύ καιρό. Και τέλος προς την Ισπανίδα ε, συνάδελφο με την οποία πολλές συνομιλίες έχουμε και τις οποίες την ευχαριστώ αλλά πραγματικό είναι θέμα το πώς θα βοηθήσουμε εκείνες τις χώρες που πλήττονται ιδιαίτερα μέσω του Frontex, μέσα στις βοήθειες ε, διοικητικής μορφής ε, για να μπορέσουν έτσι να διακανονίσουν αν θέλετε λογικά ένα μεγαλύτερο αριθμό ετούντων ασυλών και επίσης για να αποφευχθεί η οργανωμένη εγκληματικότητα όπως αυτή τη στιγμή περνάει από την Τουρκία και όπου προωθούνται 150.000 ετούντες ασύλο το χρόνο που δεν είναι πραγματική βέβαια ετούντες άσυλο αλλά που προωθούν κατά αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα. Ευχαριστώ κυρία Χέρς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πάντα νομίζω εργαστήκαμε εις βάθος στους διάφορους ορισμούς και τις διάφορους τομείς και εγώ σας ευχαριστώ για αυτά από πλευράς μου. Για μένα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η συνένωση αυτών των δύο διαφορετικών μορφών καθεστώτος, αν θέλετε, καθεστώς προστασίας. Γιατί δηλαδή, καταρχήν έχουμε το καθεστώς των προσφύγων σύμφωνα με τη της Γενέβης. Αν δούμε το κατάλογο που υπήρχε μέχρι στιγμής, Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση αν προωθείται δηλαδή το καθεστώς ε, του ετούτος άσυλο ή του πρόσφυγα. Οι ορισμένου τομεί θα ήταν καλό να έχουμε προσέγγιση των ορισμών, παραδείγματο στην πρόσβαση στην αγορά εργασία, γιατί όταν έρθει κάποιο εδώ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ε, έχει άμεση πρόσβαση στην αγορά εργασία. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, θα πρέπει να του δίνουμε τη δυνατότητα γλωσσικών γνώσεων, όπου λέμε ότι είναι άσχετο πόσο θα μείνει κάποιος και για ποιο λόγο. Παρ' αυτά είναι λογικό να έχουμε αυτές τι διαφορετικέ μορφέ, γιατί μια φορά μπορεί να υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Εάν τα άτομα αυτά αναγνωρίζουν στο μέλλον μόνο σύμφωνα με την σύμβαση για τους πρόσφυγες, ορισμένοι δεν θα εντάσσονται πια Γιατί θα πρέπει να διατηρήσουμε τις δύο αυτές μορφές. Κατά τη γνώμη μου αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι το θέμα κατά πάσα να κινηθούμε πιο πολύ προς την ε, κοινωνική πρόνοια ή προς την αγορά εργασία. Ε, βλέπουμε ότι όταν έχει κανένας πρόσβαση στην αγορά εργασία μπορεί και γλίγορα να μάθει τη γλώσσα, να μάθει τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, κράτος δικαίου κλπ παρά αν κάποιος ε, μένει με κοινωνικά επιδόματα σε κάποιο στρατόπεδο, αν θέλετε, σε κάποιο διαμέρισμα ή κάπου εκτός όμως της κοινωνίας της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν το γλυγορότερο να έχει πρόσβαση το άτομο αυτό στην αγορά εργασίας γιατί πρόκειται και για θέματα ενσωμάτωσης στην κοινωνία. Κατόπιν. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό να υπάρχει αμοιβαίο ας πούμε δικαίωμα ασύλου μέσα στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα πρέπει εμείς σαν κοινοβούλια ή κομισιόν να φροντίσουμε οι όροι αυτοί που θέλουμε να ισχύουν στον Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Όχι. Τελευταία ερώτηση δύο συναδέλφων που έχουν υποβάλει μία τροπολογία πριν δώσουμε το λόγο στον Κομισιόν και στον για να απαντήσει. Ποια είναι η άποψη της εισηγήτρια για την τροπολογία 63. για το θέμα του ε, τικού προσανατολισμού που υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση του στα διάφορα κράτη-μέλη. Εγώ ξέρω κάποιο κράτος μέλος όπου υποβάλλονται οι άνθρωποι αυτοί σε πάρα πολύ ταπεινωτικά τεστ για να αποδείξουν οι άνθρωποι αυτοί τον ε, σεξουαλικό του προσανατολισμό. Δεν θα σα πω ποια χώρα είναι και τι τεστ είναι αυτό, αλλά είναι φοβερό. Γιατί το κείμενο τη Κομισιόν είναι αδύναμο, γι' αυτό υποβάλλουμε εμεί μια άλλη τροπολογία. λέει ότι το κράτο μέλος μπορεί να ορίσει μια κοινωνική ομάδα βασιζόμενη στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Βατάσκο Γκέν, δεν ξέρω, κυρίως κύριο τι είναι. Κυρία Πρόεδρε, είχαμε εξηγήσει την πρότασή μας και προηγούμενη φορά και είχαμε σχολιάσει τις πρώτες κατευθύνσεις της εισηγήτριας. Αυτό που ελπίζουμε τώρα για το επόμενο εξάμεινο είναι να γίνουν, να σημειωθούν σημαντικές πρόοδες στο διάλογο μεταξύ των δύο συνυπευθύνων νομοθετικών οργάνων και να εγκριθεί υπό την Ουγγρική Προεδρία η οδηγία αυτή. Στο τεχνικό επίπεδο του Συμβουλίου δηλαδή υπήρξε πρόοδος και ελπίζουμε τις επόμενες εβδομάδες κάτι ανάλογο να γίνει και με τη γνωμοδότηση του ή με ως προς την ενδεικτική ψηφοφορία για να προχωρήσει ο τριμερής διάλογος και να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε αρκετά σύντομα. Στο κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ για το σχόλια αυτό. Τα σχόλια του κ. Ρομέρο Λόπες μας τόνισαν ότι είναι σημαντικό η δέσμη αυτή για το άσυλο να μπορέσει επιτέλους να εφαρμοστεί. Το θέμα δεν είναι απλώς να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη της διάσκεψη της Σύμβασης της Γενέβης αλλά να τεθεί το θέμα σοβαρής βλάβης και γι' αυτό υπάρχουν τα δύο θέματα. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει το καθεστώς του αιτητού ασύλου να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα του αιτητού και όχι στους ορισμούς ή τις μεμονωμένες ε, εξετάσεις ατομικών περιπτώσεων. Εντάξει, μιλήσαμε για θέματα υγείας και είπαμε ότι πρέπει και αυτά να είναι επίπεδου τέτοιου ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες του κάθε προσώπου και όχι να βασίζεται η νομοθεσία σε αυτά που ζητάει το ένα ή το άλλο κράτος μέλος. Για τα δικαιώματα των παιδών συμφωνούν οι σκιώδεις να συμπεριληφθούν και αυτά. Τώρα σε ποια στιγμή ακριβώς θα το δούμε, αν θα είναι στην επεξηγηματική έκθεση ή στα ίδια τα σημεία θα το δούμε. Και μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε και τη διατύπωση γιατί υπάρχουν και εδώ διαφορές μεταξύ των τροπολογιών που έχουν σχετικώς κατατεθεί. Όσο για την 104 που μιλάει για τα γλωσσικά, και αυτό είναι κάτι επί το οποίο νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί συμφωνία μεταξύ των σκιωδών. Και θα συνεννοηθούμε και με τους συντάκτες για να ξέρουν και αυτοί ακριβώς πώς έχει η τροπολογία αυτή. Για την οικογένεια τώρα εκείνη η τροπολογία, ναι γενικά συμφωνούμε και από αυτού και ως προς τους ορισμούς και ως προς τους στόχους αλλά η συμφωνία αυτή πρέπει να καλύπτει όλα τα τμήματα της δέσμης για το άσυλο. Τώρα για τα συγκεκριμένα, όπως η τροπολογία 63 ας πούμε, το κείμενο λέει ότι επειδή οι συνθήκες της χώρας προέλευσης καθορίζουν αν κάποια κοινωνική ομάδα θεωρείται εν κινδύνο ή όχι, μπορεί κάποιος που προέρχεται από τις Ηνωμένε Πολιτείες να μην θεωρηθεί το ίδιο σε κίνδυνο όπως κάποιος από την Ιαμαϊκή ως προς το σεξουαλικό του προσανατολισμό ας πούμε. Είναι θέμα δηλαδή συνθήκων στη χώρα πραέλευσης. Αν δηλαδή συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι μια χώρα προέλευσης είναι υψηλής ποιότητας ή όχι. Να αυτά για τις συγκεκριμένες μεμονωμένες περιπτώσεις αυτό για το 63. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσω επίσης με τους συντάκτες μετά όμω, μετά. Για το χρονοδιάγραμμα Καλό θα ήταν ίσως η Επιτροπή να εξετάσει τις συμβιβαστικές στη συνεδρίασή της του τέλους Ιανουαρίου, ώστε μετά το Φεβρουάριο να εγκρίνουμε αν, αν συμφωνούν και οι άλλοι βέβαια, καθώς και η παραεδρία. Καλά θα δω, θα δω λέει η Προεδρία έχει κανείς καμία σοβαρή αντίρρηση ή η γραμματεία το θεωρεί ιδιαίτερα δύσκολο αυτό το χρονοδιάγραμμα. Όχι, τότε θα ακολουθήσουμε αυτό. Θα δούμε δηλαδή τις συμβιβαστικές τέλη Ιανουαρίου και μετά την ενδεικτική ψηφοφορία αρχές Φεβρουαρίου δεν έχω τις ακριβείς ημερομηνίε, αλλά περίπου έτσι. Μάλιστα έτσι τελειώνει και αυτό το σημείο και περνάμε τώρα στο σημείο 8. Το πριν της ώρας του. Φαντάζομαι ότι έρχονται όλοι όσοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ελπίζω να συμφωνεί ο κύριος Μπουσουτήλ να αρχίσουμε αν και είναι νωρίτερα. Και ζητώ συγγνώμη γιατί στη μέση της συζήτησης αυτής θα αντικατασταθώ γιατί πρέπει να πάω σε άλλη επιτροπή. Αυτό το 8 λοιπόν αφορά την απαλλαγή του 2009, εισηγητής είναι ο κύριος Μπουσουτήλ και η Επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη 6 γνωμοδοτήσεων για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Όσοι θέλουν να φύγουν παρακαλώ να το πράξουν ηρέμως. Α, τα έχασα τώρα. Ε, μια έξι νομοδοτήσεις για την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, μία για την απαλλαγή του προϋπολογισμού της Κομισιόν και πέντε για τις πέντε υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι ελεύθερων θεμελιών δικαιωμάτων, τα κατάχρηνα κροτικών, του Urban Σύμπολ και Frontex. Και για να τα συζητήσουμε αυτά, καλέσαμε και τους διευθυντάς Επαναλαμβάνω όσοι θέλουν ιδιωτικές συζητήσεις να το κράξουν έξω. Τακ, τακ, τακ. Ευχαριστώ. Καλέσαμε λοιπόν τους διευθυντάς των πέντε υπηρεσιών για να μας κάνουν μια παρουσίαση. Ο καθένας και δεν ξέρω πόσοι έχουν καταφθάσει αλλά Καλέσαμε τον κύριο Μανολόπουλο, υπεύθυνο τη Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, τον Wolfgang Goods, διευθυντή του EMCDDA, τον κύριο Hans Garais από την Ευρωδίκ, τον αναπληρωματικό διευθυντή του ΣΥΠΟΛ και τον διευθυντή του Frontex. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Βουσουτήλ για να μας παρουσιάσει τον έγγραφο εργασίας του και θα αρχίσει μετά η συζήτηση και θα απαντήσει η Κομισιόν και οι άλλες υπηρεσίες που ανέφερα. Ο εισηγητής θα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου και η δε διορία κατάθεση τροπολογιών θα λήξει στις 3 Φεβρουαρίου. Δεν έχουμε άλλη επιλογή και η ψηφοφορία θα γίνει 28 Φεβρουαρίου. Ορίστε κύριε Βουσουτήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο εργασία μου, όπω είπατε κι εσεί, αφορά τι πέντε υπηρεσίε που είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα αλλά φορά και την Κομισιόν διότι ο προϋπολογισμός προφανώς σχετίζεται με θέματα δικαιοσύνης, ασφαλείας κλπ. Το έγγραφό μου λοιπόν είναι πολύ απλά οργανωμένο. Έχω παρουσιάσει σε δύο συναδέλφους τα κείμενα που αφορούν στο, στην ετήσια έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου την κάθε υπηρεσία και μετά την απάντηση της υπηρεσίας αυτής στο Ελληνικό Συνέδριο. Και μετά έγραψα πρόσθετα ερωτήματα με βάση τις απαντήσεις της κάθε υπηρεσίας. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ακούσω τι έχει να πει κάθε μια από αυτές τις υπηρεσίες καθώς και η Κομισιόν σαν συμπλήρωμα των δικών μου συμπληρωματικών ερωτήσεων. Για τα μέλη που δεν έχουν διαβάσει αυτό το έγγραφο εργασίας ακόμη, Ίσως θα έπρεπε να περιγράψω τα κυριότερα σημεία της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά εσείς θα μου πείτε πώς να το κάνουμε. Να ακούσουμε πρώτα τις απαντήσεις του καθενός. Α, έτσι μπορεί οι συνάδελφοι να μην καταλάβουν ποια υπηρεσία απαντάει σε ποιον. Ή μήπως θα έπρεπε πρώτα να θέσουμε τα θέματα της κάθε υπηρεσίας και να απαντάει μία-μία. Εσείς να μου πείτε. Με τα χαράς. Η δεύτερη πρόταση είναι η καλύτερη, μία-μία. Μεταξύ άλλων και διότι δεν έχει ακόμη έρθει ο εκπρόσωπος μίας από αυτές τις υπηρεσίες. Με ό,τι σειρά θέλετε αλλά ο αναπληρωματικός διευθυντής της ΥΠΟΛ δεν έχει έρθει ακόμα, σας το είπα. Όποια σειρά θέλετε λοιπόν. Ωραία. Τότε θα αρχίσω με την Κομισιόν. Α, δεν είναι ούτε Κομισιόν εδώ. Ε, τότε την Ευρωδίκ. Ήρθε η Κομισιόν. Ναι. Ήρθε τώρα βγάζει το παλτό της. Λοιπόν, μόλις βάλει και τα ακουστικά, μάλιστα μέχρι να καθίσουν λοιπόν, ας πάω στην Ευρωθήκ. Βασικά στην έκθεση του το ελληνικό Συνέδριο μας είπε ότι το 2007 και το 2008 υπήρχαν πολλές καινές θέσεις στην Ευρωδίκ. 33% και 66% αντιστοίχως. Και το 2009 δεν έγινε καμία πρόσληψη. Ερώτησα λοιπόν την Ευρωδίκη γιατί υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες στις προσλήψεις και ακόμη και με την έλλειψη αυτή προσωπικού θεωρεί ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντά της. Για την επιλογή του προσωπικού επίσης θα ήθελα να ρωτήσω την ευρωδική. Τι θα γίνει με τα συμβόλαια που είχε υπογράψει προηγουμένως, διότι το ελεγκτικό συνέδριο θεώρησε ότι μερικοί υποψήφοι είχαν επιλεχθεί με διαδικασία όχι και τόσο νόμιμη, παράτυπη. Τι θα γίνει λοιπόν με τα συμβόλαια που υπογράφτηκαν βάσει της παρατύπου διαδικασίας. Ναι, ευχαριστώ κύριε Κέλλερ, Έχεις ζητήσει το λόγο. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι για την Eurojust. Όχι τότε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Eurojust, κύριος Χάνς Γιάρβερ, ο οποίος ε, είναι εκτελεστικός διευθυντής της Eurojust. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας, λέγομαι Χάνς Γιάρεν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω το συντομότερο στις ερωτήσεις. Ρωτήσατε γιατί υπάρχουν δυσκολίες ε, για την πρόσκληση προσωπικού. Εργαζόμαστε σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο, κυρίως ε, ε, στη Χάγη και Υπάρχουν, ε, υπάρχει ένας ε, μικρός αριθμός ε, προσωρινών συμβασιούχων, δηλαδή, και κάτι τέτοιο μας έχει δυσκολεύσει στο, στο παρελθόν για να ανταγωνιστούμε. Ε, επίσης υπάρχει έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Ελπίζω να έχει ξεπεραστεί όμως αυτή η δυσκολία τώρα. Από την άλλη, μία ακόμη εξήγηση μπορεί να είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε το, ε, ε, ε, διαδικασία πρόσληψης, δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάποιες παράλληλες δραστηριότητες ε, και να βελτιώσουμε την αλληλουχία μας. Επίσης, εφαρμόζεται τώρα ε, από το 2010 το πλήρες σχέδιο πρόσληψης και επίσης ζητήθηκαν και τα τελευταία νούμερα για τις κενές θέσεις. Το 2009 είχαμε 185 θέσεις από τις οποίες το 2009 πληρώθηκαν 141, είχαμε 44 κενές θέσεις υψηλού επίπεδου. Το 2010 των 85 ε, από τις οποίες 163 έχουν πληρωθεί. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε 22 καινές θέσεις στα τέλη του 2010. Έχουμε λοιπόν 50% ε, μείωση. Τώρα η ερώτηση που τέθηκε είναι πιστεύετε ότι η Eurojust μπορεί να πληρώσει τα καθήκοντά της. Ναι, το πιστεύουμε, αλλά φυσικά θέλουμε να βελτιώσουμε τις εσωτερικές μας διαδικασίες και τις διαδικασίες πρόσληψης. Επίση, τέθηκε και ερώτηση τι θα γίνει με τις συμβάσεις που συνάφθησαν μέσω παράτυπης διαδικασίας. Πρέπει να παραδεκτώ ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει για νομικούς λόγους, γιατί αυτές οι συμβάσεις έχουν συναφθεί, έχουν περάσει και τη δοκιμαστική περίοδο οι υπάλληλοι. Έτσι λοιπόν δεν βλέπω δυνατότητα εμείς ως Γιούρτζες να κάνουμε το οτιδήποτε. Και ούτε καν βλέπουμε αναγκαιότητα για να λείψει δράση σε αυτόν τον τομέα. Ελπίζω να απάντησα πλήρως. Είστε ικανοποιημένα κύριε Σιγητά. Ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν είμαι και τόσο ικανοποιημένο με το τελικό σχόλιο, γιατί ουσιαστικά η Eurojust παραδέχτηκε εδώ ότι έχουν προσληφθεί κάποια άτομα βάσει παρατύπης διαδικασίας. Και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα η Eurojust. Επομένω και εμεί θα καταλήξουμε στα δικά μα συμπεράσματα βάσει αυτή τη απάντηση. Από την άλλη, είμαι ικανοποιημένο για την απάντηση στι πρώτε ερωτήσει. Βέβαια, αν και κάποιοι άλλοι, άλλοι βουλευτέ θέλουν ε, να θέσουν ερωτήσει στου αντίστοιχου οργανισμού, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα επανέλθω στην Κομισιόν το 2009 το επίπεδο της ε, εφαρμογής ε, των δεσμεύσεων ήταν 97,7% και αυξήθηκε λοιπόν από το 2008 και η εφαρμογή των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89,6%. Είχαμε αύξηση δηλαδή και εκεί. Όμως ε, είχαμε και αρκετή αρκετά υψηλό αριθμό κυρώσεων, 8,5%. Έτσι λοιπόν θέλω να ρωτήσω πώς ε, τα διάφορα κονδύλια και προγράμματα εφαρμόστηκαν το 2009 θα ήταν δυνατό να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το ε, ταμείο, για τις επιστροφές και για τα εξωτερικά σύνορα και πότε οι εκθέσεις ε, θα είναι διαθέσιμες ε, γιατί μας έχει υποσχεθεί τις εκθέσεις αυτές η Κομισιόν ε, και σε ό,τι φορά τώρα το ΣΥΣ 2. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς δόθηκαν τα κονδύλια, μάλλον πώς δαπανήθηκαν τα κονδύλια το 2009, τα κονδύλια που είχαν εκταμιευθεί ε, για το ΣΥΣ 2 και θέλω να ρωτήσω για τις ακυρώσεις πληρωμών, γιατί είχαμε τόσο υψηλό ποσοστό κυρώσεων πληρωμών το 2009 και ε, σε ποιες ε, γραμμές δημοσιονομικές έλαβαν χώρα αυτές οι κυρώσεις. Ε, ελπίζω να μπορεί να απαντήσει η Κομισιόν σε ερωτήσει αυτέ, γιατί τι είχαμε στείλει εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέντ. Ελπίζω να έχει καθίσει η Κομισιόν, να, να Άκουσε τις ερωτήσεις γιατί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Θέλετε να πάρετε το λόγο πριν την Κομισιόν, παρακαλώ. Θέλετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ακούσετε πρώτα την απάντηση της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Πουσουτήλ ε, θα αναφερθεί και σε άλλες υπηρεσίες. Α, μία-μία. Εντάξει, με τη σειρά. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Okay, thank you. I'm Stephanie Carillon um, Λέγομαι Στεφανή Καριών, είμαι από την Γάμα Δελτα Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει που τέθηκαν. Να κάνω μια δήλωση καταρχήν. Αν διαβάσουμε την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου, εμεί είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την έκθεση, γιατί δεν ε, φαίνεται να υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Το βλέπω αυτό και από τις δικές σας ερωτήσεις γιατί αφορούν τα ποσοστά εφαρμογής. Δεν ξέρω αν θέλετε λεπτομέρειες για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών. Μπορώ να σας πω ότι αφορά το Shared Management Fund, το ταμείο αυτό που είναι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών μας. μιλάμε για 98-99 με 100% σε ό,τι αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει σε πλήρη σχεδόν ε, εφαρμογή των ε, τεσσάρων Ταμείων Κοινή Διαχείριση. Και σε ό,τι αφορά και το Ταμείο Επιστροφή και το Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα, στο οποίο αναφερθήκατε συγκεκριμένα. Έχουμε λοιπόν καλύψει την καθυστέρηση που είχαμε το 2008. Σε ό,τι αφορά την μεσοπρόθεσμη, την ενδιάμεση αξιολόγηση, στο πρώτο ήμιση του 2011 την περιμένουμε θα τη τώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Επομένως θα το εξετάσουμε. Και κάνατε και μια ερώτηση για το ΣΥΣ 2, για το βαθμό εφαρμογής. Οι πιστώσεις πληρωμών και πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων φτάνουν στα 72-73%. Αυτό αντικατοπτρίζει το ότι είχαμε τεχνικά προβλήματα με το ΣΥΣ 2 το 2009, δεν το γνωρίζετε. Επίσης είχαμε και ένα αποθεματικό στο 4 του 2009 και φυσικά καθυστέρησαν κάποιες πληρωμές. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και τώρα το επίπεδο ακυρώσεων. 8,5%. Έχουμε 44 εκατομμύρια συνολικά. Ένα μεγάλο τμήμα αφορά συστήματα πληροφορική. Πάλι είχαμε αυτό το πρόβλημα με τα συστήματα πληροφορική. Έπρεπε να καθυστερήσουμε λοιπόν κάποιε πληρωμέ. Ένα μεγάλο τμήμα είναι οι οργανισμοί, οι υπηρεσίε. 22 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια από τη Frontex, ε, 4,5 εκατομμύρια από την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε ΠΟΛ 7 εκατομμύρια. 22 εκατομμύρια συνολικά λοιπόν πληρωμές ακυρώθηκαν από, του από τους οργανισμούς. Και έχουμε και προγράμματα που δεν λειτουργήσαν τόσο καλά όσο αναμενόταν κυρίως στην άμεση διαχείριση και στην καταπολέμηση και πρόληψη του κλίματος. Αυτά. Ελπίζω να απάντησα σε όλες σας τις ερωτήσεις. Αν έχετε κι άλλες, ευχαρίστως. Yes, thank you. Can I come back on the issue of... Ναι, μπορώ να επανέλθω στο θέμα των ακυρώσεων. Μπορούτε να επαναλάβετε το συνολικό ποσό του 8,5% πόσα εκατομμύρια ήτανε και επίσης ποιο είναι το ποσοστό του προπολογισμού σε πόλ που αντικατοπτρίζεται από τα 7 εκατομμύρια που ακυρώθηκαν. Ένα λεπτό να κάνω του υπολογισμού μου και θα σας πω. Περιμένουμε η Κομισιόν να υπολογίσει τα ποσοστά και θα εξετάσουμε τα μεταξύ και τις άλλες εκθέσεις για τις διάφορες υπηρεσίες. Εν τω μεταξύ. It was a difficult question, I think. ήταν πολύ δύσκολη αυτή η ερώτηση. Όχι, δεν έχω το αριθμητικό στοιχείο και δεν θέλω να σας δώσω κάτι το εισφαλμένο. Δεν είναι προφανές, γιατί οι ακυρώσει των πληρωμών αφορούσαν και το 2009 και το 2008. Δεν πρέπει να δούμε λοιπόν. Πρέπει να τα υπολογίσω αυτά και να σας τα πω. Κύριε ευχαριστώ. Μήπω μπορώ να ρωτήσω ότι η Κομισιόν και τι Υπηρεσίε που εκπροσωπούνται εδώ να μα στείλουν, ε, στείλουν γραπτά τι απαντήσει, στις ερωτήσει που είπε, βάλαμε γραπτά. Έτσι όλοι οι συνάδελφοι θα έχουν στα χέρια του. Τι απαντήσει. και λόγω του περιορισμένου του χρόνου που έχουμε δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τα πάντα αυτή τη στιγμή και θα ήταν κρίμα να μην πάρουμε απαντήσεις όλα. Για να περάσουμε τώρα στις άλλες υπηρεσίες, στο Οργανισμό Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και ε, ε, του Εθισμού. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι μετέφερε 339.000 ευρώ από ε, τα χρήματα που προβλέπονται το 2009 για τις διοικητικές δαπάνες, 26% δηλαδή. Και θα ήθελα να ρωτήσω την υπηρεσία αυτή τι έκανε για να βελτιώσει τον προγραμματισμό του για να μπορέσει να χρησιμοποιεί τον προπολογισμό του πιο αποτελεσματικά. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω το κέντρο αυτό Εν των χρημάτων που επιστρέφθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μετάφρασης ερωτώ εδώ την Κομισιόν επιβεβαίωσε η Κομισιόν ότι αυτό τα χρήματα ε, θεωρούνται δεδομένο εισόδημα και κατά πόσον υπάρχουν συμπληρωματικές, ε, συμπληρωματικά μέτρα για να υπάρχει καλύτερη σαφήνεια. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πρωτού προχωρήσουμε, θα ρωτήσω το υπόλοιπο μέλη αν έχουν κάποιες ερωτήσεις. Πριν ζητήσουμε από την υπηρεσία να απαντήσει. Όχι, ωραία. Λοιπόν, ο τον διευθυντή αυτού του, της υπηρεσίας του EMCDDA να απαντήσει και με τα Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν όσον αφορά τις ερωτήσεις για την μεταφορά αυτήν του διοικητικού ε, από το διοικητικό προπολισμό το 339.000 που είναι το 2% του ε, προπολογισμού μας όχι 26% του συνολικού μας προπολογισμού, αλλά 2%. Και μέσα 339.000 αυτές τα 26% είναι καθαρό διοικητικό χρήμα. Και το υπόλοιπο 74% αφορά τη μετακόμιση στο νέο κτίριο όπου εκεί είμαστε θύματα διαφόρων ε, καθυστερήσεων που οφείλονται στον ε, νοικοκυριακή και η μεταφορά έγινε πολύ πιο αργότερα από ό,τι προβλέπαμε. Και οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται στον ιδιοκτήτη του κτηρίου που είναι οι λιμενικές αρχές της Πορτογαλίας. Βελτιώσαμε όμως, διευκρινίσαμε τις ε, ε οδηγίες μας προς τους συναδέλφους που εργάζονται για, την, για τον έλεγχο του προπολογισμού και για το λογιστικά για να μπορέσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον κάτι τέτοιο. Υπήρχαν και πέντε συγκεκριμένες ε, συγκεκριμένα μαθήματα προσανατολισμού για τα άτομα αυτά και ενημέρωση των μελών για τη βελτίωση των, της διαδικασίας ενημέρωσης κλπ. Και όλα αυτά εντάσσονται σε αυτόν τον προπολογισμό. Για το άλλο θέμα τώρα, που αφορά το εσωτερικό έσοδο, με τα χρήματα αυτά που επιστρέφησαν από το κέντρο μετάφρασης, γιατί τελικά το κόστος ανασελίδα για το κέντρο ε, μετάφρασης ήταν χαμηλότερο από ό,τι προβλέπετο και γι' αυτό μειώθηκε το κόστος. Αυτά τα χρήματα θεωρούνται χρήματα εσωτερικού εισόδων. Αυτή η άποψη βασίζεται στον δημοσιονομικό προβλησμό που αναφέρεται στην επανάκτηση ποσών που έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί η Κομισιόν έχει μία, έναν ορισμό του θέματος που δεν αναφέρεται στα εσφαλμένα καταβεβληθέντα χρήματα αλλά και σε αλλαγές που εμφανίζονται αργότερα. Γιατί εδώ είχαμε μια εκτίμηση προεπολισμού από το κέντρο μετάφραση και μετά αποδείχθηκε ότι ήταν χαμηλό το κόστος και μας επιστρέψανε τα χρήματα αυτά και αυτό δεν αφορά μόνο τη δική μας υπηρεσία αλλά και πολλές άλλες. Και γι' αυτό θα ήταν καλό να δούμε ποια είναι η οριζόντια προσέγγιση του θέματος αυτού, αν είναι πρόβλημα. Αμφιβάλλω, μέχρι στιγμή δεν υπήρχε αντίδραση Κομισιόν για το θέμα αυτό. Θα μπορούσα να φανταστώ όμως ότι η Κομισιόν θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό μέσα στα πλαίσια της ε, επερχόμενης ε, αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου κανονισμού για τις υπηρεσίες. Άλλο τίποτα δεν έχω να πω, αν θέλει και άλλες ερωτήσεις να σα απαντήσω. Ευχαριστώ κύριε που σου το λέει. από την απάντηση αυτή. Κύριε Μασκάλα. Θα μπορούσα να μας πει η Κομισιόν κατά πόσο θα επιβεβαιώσουν την άποψη των υπηρεσιών σε αυτό ή όχι. Θέλω σε ευχαριστώ. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Μάλιστα. Αυτό το θέμα τέθη από διάφορες υπηρεσίες. Από ό,τι φαίνεται έχει δίκιο το ελληνικό συνέδριο και θα φροντίσουμε την επόμενη φορά να υπάρχει σωστή ταξινόμηση. Θα έπρεπε να υπάρχει σε διάφορα εισοδήματα. Και έχει μπει τώρα στα άλλα εισοδήματα, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ. Να περάσουμε στην επόμενη υπηρεσία. Ναι, ναι, να περάσουμε. Frontex. Και να αρχίσω υποβάλλοντας ε, ερωτήσει στη μεταφορά από το προπολογισμό 2009. Γιατί υπήρχαν τόσες πολλές μεταφορές και ακυρώσεις το 2009. Ποιο ήταν το τμήμα του προπολογισμού της υπηρεσίας που επλήγει από αυτό. Πώς βελτίωσε η υπηρεσία αυτή τις προσπάθειες από τότε. Ποια είναι τα μέτρα που ανέλαβε Αυτές οι προσπάθειες έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Στην επερχόμενη μεταρρύθμιση, ε, αναθεώρηση συγγνώμη της υπηρεσίας του Frontex. Αυτά. Before we ask for the answer, I would like to ask whether there is somebody else who would like to... Madam Keller, please. Κανείς άλλος. ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω μήπως με βάση αυτές τις χρηματικές μεταφορές από χρόνο σε χρόνο θεωρείτε ότι απορροφήθηκαν όλα αυτά ή μήπως έμεινε πλεόνασμα. Οι δε κενές θέσεις, οι χειρεύουσες δηλαδή, μπορούν να πληρωθούν ίσως με το υπάρχον προσωπικό. Άλλο. Ναι. Σε ποιους τομείς της δραστηριότητας του Frontex έγιναν οι περισσότερες μεταφορές το 9. Δεύτερον, νομίζετε ότι ο προϋπολογισμός σας είναι υπερβολικά υψηλός και πρέπει να μειωθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτε άλλο. Ο Μαγέρ. Εκτάζουμε, και εκτός μικροφώνου. Εγώ θα αντίστροφη ερώτηση, γιατί τώρα που για πρώτη φορά ε, ζητήθη έντονη βοήθεια του Frontex ε, στην Ελλάδα, κατά πόσον έχει αυξηθεί το κόστος προσωπικού από τούτο το έτος, από τούτο που χρησιμοποιούν δηλαδή στην Ελλάδα και κατά πόσον στα πλαίσια αυτά θα χρειαστούν περισσότερα άτομα και χρήματα μια που το έργο τους στα ελληνοτουρκικά σύνορα είναι πολύ πιο έντονο από ό,τι είχε προβλεφθεί. I would like Α, ωραία. Τότε ο εκπρόσωπος του Πρόντεξ για να απαντήσει. Μάλιστα, Καλησπέρα σας. Ε, πράγματι, οι πολλές μεταφορές και ακυρώσεις ήταν κάτι που διαπιστώσαμε και εμείς στη χρήση του προϋπολογισμού μας και τη διαχείρισή μας. Υπάρχει εδώ ολόκληρο ιστορικό, δεν, είναι η πρώτη φορά που συζητούμε για αυτό το θέμα. Θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως αν μου δίνατε την άδεια να απαντήσω λεπτομερώς στα ερωτήματα του κύριου Βουσουτήλ, αλλά αυτό θα το κάνω αργότερα και τώρα θα απαντήσω μόνο στα ερωτήματα που μου τέθηκαν τώρα. Πρώτον, για τις μεταφορές ε, που είναι και τα σημεία του προπολογισμού μας που μας έθεσαν το περισσότερο πρόβλημα. Οι κύριες τρεις είναι οι κοινέ θαλάσσιες επιχειρήσεις, δεύτερον η επιμόρφωση και τρίτον το ICT που λέμε που είναι προγράμματα χαρακτηριστικά για μια τέτοια υπηρεσία. Αυτοί οι τρεις τομείς λοιπόν, ιδίως το ICT όμως, ε. Αλλά δεν είναι πρώτη φορά, το είπα και πέρυσι. Αν περιοριστούμε σε ένα έτος, κατανοούμε εύκολα ότι πρέπει να σεβαστούμε τον ενιάφσιον χαρακτήρα του προϋπολογισμού, αλλά για τη χρήση του προϋπολογισμού του 9, τώρα μόνο έχουμε τους τελικούς αριθμούς. Μπορεί να είναι καθυστερημένοι, αλλά τώρα έρχονται. 91% ήταν οι πληρωμές η απορρόφηση των πληρωμών περίπου το ίδιο με τον προηγούμενο χρόνο δηλαδή του 8 και και οι υποθέσεις που κάνουμε για τις ε, δεσμεύσεις ήταν 80% πολύ καλύτερες από τον προηγούμενο χρόνο αλλά οι αριθμοί αυτοί δεν είναι ακόμη τελικοί ούτε ανταποκρίνονται στους στόχους που είχαμε καθορίσει και μόνοι μας εξάλλου. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι εδώ μιλάμε για επιχειρήσεις όπου η κατάσταση αλλάζει ζωτικά και γρήγορα. Μιλάμε για τη χρήση του 9 βέβαια, αλλά αν πάρουμε για παράδειγμα το 10 θα δούμε ότι συνέβησαν δύο μεγάλες αλλαγές. Δραστική μεταφορά από θαλάσσια σύνορα σε χερσαία ιδίως μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο ακριβό να εφαρμόσει κανείς κοινέ θαλάσσιες επιχειρήσεις με ελικόπτερα και τέτοια παρά με χερσέ, για χερσές όπου χρησιμοποιούμε οχήματα, σκύλους, σκύλες και είναι πιο ακριβό αυτό και για να τα σχεδιάσουμε όλα αυτά για διάρκεια μεγαλύτερη από ένα χρόνο πριν συμβούν είναι δύσκολο, έχουμε 27 χώρες να συντονίσουμε και οι αναλύσεις που κάνουμε δεν μπορούν να είναι ακριβέστατες εκ των προτέρων. Έχουμε και τους εταίρους μας στο Σέγγεν και λοιπά όλα αυτά. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Για το δεύτερο ερώτημα τώρα, για το επίπεδο του προϋπολογισμού. Δεν πρέπει να διαχωρίσουμε το δικό μας προϋπολογισμό μόνο από τους υπόλοιπους. Πρέπει όλο το τρίγωνο να δούμε, δηλαδή δημοσιονομικούς πόρους, ανθρώπινους πόρους, που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας και τρίτον, τρίτη γωνία του τριγώνου, η θέληση και δυνατότητα των χωρών μελών να συνεργαστούν. Εδώ είναι θέματα θέλησης όλα αυτά, θέλησης. Δεν υπάρχει τρόπος να υποχρεώσουμε τις χώρες μέλη εκτός από τις ομάδες βέβαια με παρέμβαση στα σύνορα δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε εκτός από είναι λοιπόν πολύ πολύ πλοκά όλα αυτά και δεν θα έλεγα βέβαια ότι είναι πολύ ψηλός ο προπολογισμό μας γιατί αντίθετα υπάρχει ακόμη λόγος να αυξηθεί ο προπολογισμό ιδιαίτερα φέτος και του χρόνου και τα άλλα επόμενα χρόνια. Το κυριότερο θέμα για τους πόρους είναι οι ανθρώπινοι πόροι. Για να καταλάβουμε τη σημασία που έχουν οι δικταϊκές δαπάνες και οι επιχειρησιακές δαπάνες, θα σας έλεγα ότι πέρυσι 35% ήταν οι δαπάνες για τη λειτουργία, ενώ πέρυσι κάπως καλύτερα αυτό βέβαια δεν δείχνει κατά πόσον είναι σημαντικές οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουμε ή όχι, γιατί το μεγαλύτερο τμήμα του προσωπικού μας εργάζεται για τα επιχειρησιακά. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Μην το ξεχνάτε. Και τρίτον ερώτημα, αν αυξήθηκαν οι νέες δραστηριότητες αν και δεν αφορά αυτό βέβαια τη χρήση του προλογισμού του 9 αληθεύει ότι όλες οι προσπάθειες και δραστηριότητες μας από τα μέσα Οκτωβρίου πέρυσι μέχρι τώρα βασίζονται κυρίως στις ομάδες άμεσης παρέμβασης στα σύνορα. Αυτές έχουν αυξηθεί πολύ. Σημειώθηκαν μερικές καθυστερήσεις στη διαχείριση των λογαριασμών μας για τις επιχειρήσεις αυτές που είναι κατεπήγοντα ως χαρακτήρα αλλά καταφέραμε παρόλα αυτά να να επαναχρησιμοποιήσουμε το προσωπικό μας με άλλο τρόπο στις διοικητικές και άλλες επιχειρήσεις και αυτό μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις το χρονοδιάγραμμα και το κατά πόσον θα λήξουν οι επιχειρήσεις αυτές επιτυχώς γρήγορα. Η ανάλυση κινδύνου είναι κάτι που που αφορά και αυτό τον προϋπολογισμό και το σχεδιασμό και προσχεδιασμό του. Ο κυριότερος παράγοντας είναι αν οι επιχειρήσεις επιτήρησης μπορούν να περιοριστούν στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό ή αν χρειαστεί και τίποτα πρόσθετο. Για να συνοψίσω λοιπόν, το ελεκτικό συνέδριο και ο εισηγητής έχουν δίκιο σε αυτά που λένε, είναι γεγονότα αυτά που αναφέρουν, δεν κρυβόμαστε καθόλου αλλά κάναμε πολλές προσπάθειες απλοποίησης της διαχείρισης του προϋπολογισμού μας και των δομών του ώστε το Frontex να είναι πιο διαφανές αλλά δεν φτάσαμε ακόμη στο επίπεδο που θα μας επέτρεπε να πούμε ότι πετύχαμε όλους μας τους στόχους. Θετική είναι η τάση αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε ικανοποιητικό επίπεδο επίτευξης των στόχων που και εμείς οι ίδιοι είχαμε θέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρόσθετες ερωτήσεις. Ναι, θέλω κάποιες ε, διευκρινήσεις από τον κύριο Λάκιν ε, για δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το σημείο 14 στο γραφείο εργασίας Έχουμε το σχολείο του συνεδρίου ότι από τα 25 εκατομμύρια ευρώ των επιστοσιών επιχειρήσεων για τον τίτλο 3 το 2009 3,4 εκατομμύρια ευρώ που σχετίζονται με επιχειρήσεις που δεν ε, έλειξαν. Έτσι λοιπόν θέλω μια διευκρίνηση εδώ στο γιατί έγινε κάτι τέτοιο και για τη Frontex και θέλω μια συγκεκριμένη διευκρίνηση για το σημείο 17. Εδώ το ελεκτικό συνεδρίο μας λέει πάνω από 28 εκατομμύρια ευρώ το 2009 καταβλήθηκαν βάσει των μονομερών αποφάσεων επιχορηγήσεις που υπογράφηκαν από τον οργανισμό. Και αν καταλαβαίνω καλά, θεωρεί το ελεκτικό συνέδριο ότι αυτό δεν συνάδει με το σχετικό κανονισμό. Θέλω επίσης λοιπόν κάποιες εξηγήσει από τον οργανισμό εδώ για αυτό το νέο νομική μορφή συμφωνίας που ισχυρίζεται ο οργανισμός ότι ισχύει σήμερα και καλύπτεται όλες οι επιχορηγήσεις από αυτή τη συμφωνία. Πρόεδρος, πριν να ζητήσουμε από τον κύριο Λεντίνο να επανέλθει, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα για το θέμα του επίπεδου των προσλήψεων. Πιστεύετε ότι η Frontex ε, με το προσωπικό που έχει σήμερα μπορεί να επιτελέσει επαρκώ τα καθηκοντά τη. Για πρώτη φορά έχουμε αυτή την επιχείρηση Rabbit στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, πιστεύετε, καθώς ε, έχουμε και αυτή την επιχείρηση επαρκή το προσωπικό για να επιτελέσει αυτές τις δραστηριότητες. Κύριε Ματιού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω τον διευθυντή της Frontex ε, πώς σκοπεύει να βελτιώσει το συντονισμό με τα κράτη-μέλη. για να έχουμε και καλύτερη εφαρμογή του προπολογισμού, αλλά και πιο αποτελεσματική δράση επιτόπου. <clears throat> ναι, ευχαριστώ. Υπάρχουν λοιπόν ουσιαστικέ ερωτήσει εδώ που τέθηκαν. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο για να απαντήσετε και κατόπιν κομισιόν. Ευχαριστώ. σε ό,τι αφορά την ερώτηση 14α. Για αυτά τα 3 εκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να έχουν αποδεσμευτεί. Ο λόγος που δεν έγινε ήταν λόγω έλλειψης ε, κουράγιου. Υπήρχαν κάποια κρεμή ζητήματα όταν ε, έλυγε η χρήση το οικονομικό έτος και δεν ήμασταν σίγουροι αν έπρεπε να αναλάβουμε κάποιες δράσεις ή όχι. Πέρσι ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση. Έτσι λοιπόν εκεί θέλαμε να είμαστε σίγουροι. Γι' αυτό δεν έγινε αυτή η αποδέσμευση. Τώρα το δεύτερο θέμα για τη μονομερή απόφαση επιχορηγήσεων. Υπάρχει ένα ιστορικό. Άλλαξε κάποια στιγμή ο χρηματοοικονομικός κανονισμός πριν κάποιο καιρό και υπήρχε δυνατότητα οι επιχορηγήσεις ε, να δίνονται βάσει μόνο της ε, μονομερούς απόφασης ε, του φορέα που παρέχει τις επιδοτήσεις. Στην περίπτωση αυτή θεωρήσαμε ότι είναι κανόνας ε, η Frontex, ε, οι οργανώσει τη αστυνομία, η εκτοφυλακή και τα λοιπά οργανισμοί τη αστυνομία, εντό και η αξιοπιστία αυτών των οργανισμών κατά κάποιο τρόπο διαφέρει. Αν το συγκρίνουμε με την αξιοπιστία των ιδιωτικών φορέων που λαμβάνουν επιχορηγήσει από του ευρωπαϊκού οργανισμού τα ευρωπαϊκά όργανα. Το ελεκτικό συνέδριο το τόνισε αυτό το θέμα και ορθώς επισήμανε ήταν κάθετη από αυτού και εμείς επίσης ακολουθήσαμε την ίδια λογική για να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα γιατί η ερμηνεία που είχαμε στο παρελθόν δεν συνέπει με αυτή του ελεκτικού συνεδρίου η ερμηνεία του χρηματοοικονομικού έτσι λοιπόν αλλάξαμε την εσωτερική μας διαδικασία αμέσως μόλις το συνειδητοποίησαμε αυτό. Είχαμε λοιπόν μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο οπότε βασιζόμασταν στη δική μας ερμηνεία του χρηματοοικονομικού κανονισμού και αρχίσαμε να δίνουμε τις επιχορηγήσεις βάσει αυτής της μονομερούς απόφασης. Συγγνώμη που δεν κατάλαβα τη ρώτησε η κυρία Κέλλερ την πρώτη φορά για το αν αρκεί το προσωπικό ή όχι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό οργανισμό ή ε, ίδρυμα που θα έλεγε ότι <laughs> έχει επαρκέ προσωπικό. Κατανοούμε και τα δημοσιονομικά δεδομένα αυτή τη στιγμή, αλλά αν δείτε την πρόταση που υποβάλαμε και την πρόταση που υπέβαλε το Συμβούλιο της Frontex, το Διοικητικό Συμβούλιο της Frontex, για φέτος, για τα επόμενα έτη, χρειαζόμασταν 26 ε, νέες θέσεις. Όνειρο μάλλον θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε τώρα. Πάντως ε, είμαστε ελλειπήσει σε προσωπικό και πρέπει να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί σε ό,τι αφορά την ποσότητα αλλά και την ποιότητα και τον όγκο των επιχειρησιών μας. Βάζουμε τα δυνατά μας, έχουμε θέσει προτεραιότητες στις δραστηριότητές μας, αλλά φυσικά πρέπει να καταγραφεί αυτό, ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν έτσι όπως είχαν σχεδιαστεί. Για να είμαι σαφή ε, υπάρχει συμφόρηση. Τώρα, τελευταία ερώτηση για το πώ θα βελτιωθεί η κατάσταση. Για πάνω από δύο χρόνια είχαμε ένα σύστημα το οποίο ήταν επαχθές αλλά ήταν αποτελεσματικό σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των κρατών μελών και τις συνδεδομένες χώρες έγκαινη στο σχεδιασμό και σε επιχειρησιακό και σε δικαιωτικό επίπεδο. Είχαμε τις ε, διμερείς συζητήσεις ετησίως ε, όπου απευθυνόμαστε στα κράτη-μέλη του δίναμε κάποιε προθεσμίε για να μα δώσουν απαντήσει, να μα εκφράσουν τι προσδοκίε του και να μα πούν ε, σε ποιε δραστηριότητε και επιχειρήσει ε, είναι σε θέση να συμμετέχουν τα επόμενα έτη. Αυτό είναι το ένα τμήμα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ακρίβεια του προπολογισμού και το συνεχέ ε, πρόβλημα του over budgeting, του να έχουμε πλεονάζον προπολογισμό δηλαδή. Τώρα, αν εξετάσαμε το θέμα του καταλόγου AMC Αφορά τις δαπάνες για τον εξοπλισμό για κάποιες δραστηριότητες στα χερσαία και στα θαλάσσια σύνορα. Και αυτό αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό. Δηλαδή να δούμε, παραδείγματο χάρη, πόσο κοστίζουν οι περιπολίες των ελικόπτερών μας ή των διάφορων σκαφών. Έτσι αρχίζουμε να υπολογίζουμε τον προπολογισμό. Τώρα έχουμε πιο σαφείς κανόνες και πιο κατανοητούς κανόνες για τα κράτη-μέλη και για τον οργανισμό και είμαστε σε θέση να πιστεύουμε ότι είμαστε πιο ακριβείς όταν σχεδιάζουμε τις επιχειρήσεις. Και επίση ε, έχουμε προβεί και σε streamlining της υποβολής εκθέσεων Έχουμε ε, ε, επίσης δεν κλείνουμε τα μάτια μας στην αρχή του χρόνου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου για τις ε, κοινέ επιχειρήσεις. Προσπαθήσαμε να διαιρέσουμε αυτές τις επιχειρήσεις σε μικρότερες περιόδους. Και έτσι είμαστε πιο αξιόπιστοι σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την απάντηση. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε. μας ζητήθηκε και γραπτός να υποβάλλονται οι ερωτήσεις πριν την τελική διορία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τώρα θα ήθελα να φτάσουμε στο ΣΕΠΟΛ, αν είναι εδώ οι εκπρόσωποι του, γιατί σε αυτή την υπηρεσία έχω τα πιο πολλές απορίες. Πρώτον, το συνέδριο μας είπε ότι ως προς τις προμήθειες σε τέσσερις περιπτώσεις αγοράστηκαν αγαθά και υπηρεσίες χωρίς συμβόλαιο ή διαγωνισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντική δήλωση του συνεδρίου. Χωρίς συμβόλαιο ή διαγωνισμό. Και σε μια άλλη περίπτωση τη διαδικασία τη χειρίστηκε ένα μέρος του προσωπικού που δεν ήταν ειδικευμένο στις προμήθειες και γι' αυτό δεν είχε καθοριστεί, προκαθοριστεί τίποτα, δεν έγινε προσφορά ούτε Αποτίμηση. Ερωτώ λοιπόν, έγινε καμία έρευνα ως προς το γιατί αυτές οι προμήθειες δεν έγιναν νομοτύπος. Ζητήθηκε καμία ευθύνη για αυτές τις σοβαρές ελλείψεις και το νέο σύστημα που θεωρεί ότι εφάρμοσε δηλαδή τον ειδικό αξιωματούχο για τις προμήθειες λειτουργεί καλά θα ήθελα οπωσδήποτε απαντήσεις τώρα. Ναι, αλλά προηγουμένως κι άλλο ερώτημα. Στο... Έχω κι εγώ ερωτήσεις. Αλλά μήπως ήθελε ο κύριος τη Λαφτίν συγκεκριμένα την πρώτη να απαντηθεί και μετά. Ναι. Κυρία Ματιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. La Cour 900.000 ευρώ διαβάσαμε από την έκθεση του συνεδρίου ότι υπήρχαν προβληματικά αλλά λύθηκε λέει το πρόβλημα. Πώς λύθηκε, υπήρχε καμία καθυστέρηση πληρωμών από το 8 ή τίποτε άλλο. Και πώς θα απορροφηθεί αυτό το έλλειμμα, πότε θα μπορέσει επιτέλους η υπηρεσία αυτή να σεβαστεί τον ετήσιο χαρακτήρα του προπολογισμού. Για το 2008 το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι είναι προβληματικό το 30% του προπολογισμού αυτού και θεωρεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν είναι ανεπαρκή. Όσο για τη χρήση του 9, 43% του προπολογισμού έχουν αναπληθεί από το Μάρτιο του 10 εβδομαδιαία γίνονται συνεδριάσεις για τη διαχείριση από την υπηρεσία αυτή για να διευκολυνθεί ο δημοσιονομικός λέει έλεγχο. Αλλά αρνήθηκαν πάλι την απαλλαγή και πρέπει επομένω να γίνουν πολλές ακόμη αλλαγές. Μπορείτε να μας περιγράψετε σύντομα ποια είναι η δημοσιονομική κατάσταση της υπηρεσίας. Γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε το ο προϋπολογισμός αυτός 128 εκατομμυρίων να δεν μπορώ να ξαναπώ τον αριθμό είναι μεγάλος να τύχει τόσο κακής διαχείρισης επί τόσα πολλά χρόνια και πώς σκοπεύει το ΣΕΠΟΛ να τα διορθώσει όλα αυτά ευχαριστούμε πολύ θα λάβει το λόγο ο εκπρόσωπος σύντομα όμως γιατί ο χρόνος περνάει αν δεν απατώμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Πρώτα μία γενική δήλωση. Η διαχείρισή μας δεν σκοπεύει να διορθώσει λάθη του παρελθόντος μόνο. Έχουν συμβεί λάθη στο παρελθόν, αλλά ο σκοπός είναι το μέλλον. Θα επανέλθουμε μεν σε αυτό, πρώτα όμως θα απαντήσω στα ερωτήματα που θέσατε. Για τις προμήθειες, μάλιστα, υπήρξαν τέσσερις περιπτώσεις όπου οι αγορές υπηρεσιών έγιναν χωρίς την νομότυπη διαδικασία. Μία δε έγινε από κάποιον που δεν είχε τα προσόντα για να την κάνει. Το 9 όμως ιδρύθηκε η θέση του υπευθύνου προμηθειών και όλοι όσοι ασχολούνται με τις προμήθειες είναι ειδικά εκπαιδευμένοι. Ο τελευταίος εσωτερικός δημοσιονομικός μας έλεγχος έδειξε ότι όλα πάνε καλά. Είπατε αν έγινε καμία έρευνα για τα λάθη του παρελθόντος. Σας είπα και πριν και το ξαναλέω ότι δεν επενδύουμε στο παρελθόν. Δεν κάναμε μελέτες. Γιατί εμείς αυτό που θέλουμε είναι να βελτιωθεί η τωρινή κατάσταση. Όσο για την λογοδοσία, ειδικά για τις προμήθειες, δεν καθορίσαμε ευθύνες. Δεν προσπαθήσαμε να καταστήσουμε κάποιον υπεύθυνο αλλά ήδη ζητήσαμε αποζημίωση από έναν προηγούμενο διευθυντή ο οποίος θα αναλάβει τις ευθύνες του και θα πληρώσει τμήμα των χρημάτων που κατεχράστη από τους φορολογουμένους και τώρα θα σας μιλήσει ο υπεύθυνος της δημοσιονομικής μας υπηρεσίας. Χαίρετε. <laughs> Για τις μεταφορές. Φέτος εφαρμόσαμε μια διαδικασία που συνοδευόταν από ένα σημείωμα και έτσι μπορέσαμε να αποδεσμεύσουμε 900.000 άχρηστων πλέον κονδυλίων για το γάμα 8 και γάμα 9 ή ε, γάμα 1. Αυτό θα το κάνουμε και το χρόνο. Τι άλλο να σας πω. Έχουμε μια ολόκληρη επιτροπή επιτήρησης της διαχείρισης. Έχουμε συνάψει συμφωνίες που μας επιτρέπουν επίσης καλύτερη με τα επιτήρηση των πληρωμών και όπως είπε και η κυρία Ματθαίου, έχουμε εβδομαδιαίες συναντήσεις για τη διαχείριση με αναφορά. απορρόφησης του προπολογισμού. Γιατί το 9 έγιναν τόσο πολλές μεταφορές. Ο μόνος λόγος που μπορώ να βρω είναι ότι είναι ότι έγιναν όλα αυτά πριν έρθω. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτε πρόσθετο. Ορίστε εσείς εκεί κάτω. Θέλω μια αποσαφήνιση. Δεν εξηγήθηκε λοιπόν τι έγινε το 9, αλλά μας είπαν οι καινούργοι υπεύθυνη ότι προβλέπεται διαδικασία αποζημίωσης από τον προηγούμενο διευθυντή των χρημάτων του φορολογουμένου και της φορολογουμένης. Υπάρχει καμία τέτοια διαδικασία που να προβλέπει με σαφές νομικό υπόβαθρο πώς ακριβώς θα αποφεύγονται τέτοια προβλήματα δεύτερον. η, τα συμβόλαια με συμβούλους που έχετε υπογράψει και που είναι όλα παράτυπα σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο τι θα γίνουν διότι ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Τα συμβόλαια αυτά λοιπόν τα παράτυπα τι θα γίνουν, ποιο καθεστώς έχουν. Επιπρόσθετα από τις ερωτήσεις του γραπτού κειμένου θέτω. Πρώτον, εφόσον στην απαλλαγή του 8 για το 7 είχαν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, γιατί για δεύτερη συνεχή φορά έχουμε τέτοια τα ίδια προβλήματα. Γιατί δεν έγινε νωρίτερα κάποια βελτίωση, όπως λέτε ότι κάνατε τώρα. Γιατί όχι από το 8. Έπειτα, τα προβλήματα ιδιωτικής χρήσης χρημάτων ήταν από το 7 πολλές περιπτώσεις και δεν έγινε τίποτα για να αντιμετωπιστούν. Το 8 και το 9 δεν φάνηκε κάτι τέτοιο, αλλά δεν αντιμετωπίστηκε το προηγούμενο πρόβλημα. Είπατε ότι μία ή δύο, ένα-δύο μήνες πριν ορίσατε τον ειδικό ελεγκτή, επομένω τον εμπειρογνώμονα μάλλον. Για πρώτη φορά πριν από δύο μήνες λοιπόν κάνατε την παραμικρότερη έρευνα για όλα αυτά και για τις προμήθειες και για όλα και τέλος Ποιος έγραψε το εγχειρίδιο προμηθειών, αυτός ο εμπειρογνώμονας, κάποιος άλλος εμπειρογνώμονας ή κανένας που τον γνωρίζατε προσωπικά. Η κυρία Ματθέου και μετά ο κύριος Μπουσουτήλ. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς ε, συνεδριάζετε με την κυβέρνηση, δηλαδή Υπάρχει τροποποίηση, έχει αλλάξει ο τρόπος εργασίας ε, μεταξύ των διευθυντών και του ε, Governing Board. Ε, Τι υπήρξε η άρνηση της απαλλαγής από το Κοινοβούλιο. Η συνεργάζεστε πιο στενά με το Governing Board, με αυτό το Συμβούλιο το Διοικητικό. ποια σχέση έχετε, θα ήθελα να μας τα όλα αυτά. Ευχαριστώ, ο κύριος Μπουσουτήλ. Τα περισσότερα ερωτήματα που θέλω να θέσω τέθηκαν από του συναδέλφους ήδη. Πολύ ωραία λοιπόν. Πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα όμω ένα ερώτημα που δεν τέθηκε και θέλω να το θέσω εγώ. Έχει να κάνει με το σημείο 2 στο έγγραφο εργασίας. Ε, το ελεκτικό συνεδρίο μα είπε ότι όπως έχει σημειώσει ήδη στην έκθεσή του για το 2008 και τη χρήση του 8, οι δαπάνε για την οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα ε, της ΕΠΟΛ. Το Ελεκτικό Συνέδριο είπε ότι για το 2009 ο έλεγχος αυτές της δαπάνης αποκάλυψε σοβαρές λήψεις και πάλι αυτή είναι πολύ καταδικαστική δήλωση από το λεκτικό συνέδριο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, τα προβλήματα γιατί επαναλήφθηκαν το 2009, τα προβλήματα του 2008, γιατί επαναλήφθηκαν το 2009. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν για την προσωπική λογοδοσία. Ελέγξαμε προσωπικά και ε, ο πρώην διευθυντής ε, είναι προσωπικά υπεύθυνος και καταλήξαμε στο ότι υπάρχει καθαρή προσωπική ευθύνη και νομική ευθύνη. Ε, έχουμε, το χάρη, μια διαταγή για 2.200 ευρώ για ε, κάποιες ε, υπηρεσίες. Ε, αλλά πρέπει να ελέγξουμε ότι αν υπάρχει και προσωπική ευθύνη ε, του αρμοδίου υπαλλήλου που έδωσε την εντολή. Το ελέγξαμε αυτό προσωπικά και θέσαμε την ε, απέτηση αυτή έναντι του πρώην διευθυντή. Και αν υπάρχει δυνατότητα τέτοιο θέμα και σε άλλους τομείς, να είστε σίγουροι ότι θα το, πράξουμε. Θα κάνουμε τους ελεγχούς. Τώρα, για το παλιό σύστημα της συμβάσης με τους εμπειρογνώμονες κατάρτισης. Εμείς ε, αναπτύξαμε κοινά προγράμματα με τα κράτη-μέλη για ε, την εκπαίδευση των αστυνομικών ακαδημιών στην Ευρώπη. Υπήρχαμε, υπήρχαν συμβάσεις μεταξύ της ΕΠΟΛ και των αστυνομικών ακαδημιών στα κράτη-μέλη και αυτός ήταν ένας λανθασμένος τρόπος, μια λάθος προσέγγιση, το αλλάξαμε. Τώρα, το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο, στην τελευταία συνάντηση, στις αρχές Δεκεμβρίου του 10, αλλάξαμε ολοκληρωτικά αυτή την προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν ε, περαιτέρω τέτοιες συμβάσεις όπως το παρελθόν και θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι οι συμβάσεις ήδη σταμάτησαν τον Ιούνιο του 2009. Έτσι λοιπόν από τότε δεν ε, εφαρμόστηκαν ούτε εκτελέστηκαν τέτοιες συμβάσεις και τώρα θα έχουμε ε, ένα σύστημα ε, συμφωνιών επιχορήγησης. Δεν θα υπάρχουν στο μέλλον παρόμοιες συμβάσεις. Τώρα έχουμε αλλάξει και το χρηματοοικονομικό κανονισμό της ε, ΣΕΠΟΛ. Ε, διαγράψαμε μία παράγραφο ε, στην οποία μας ασκήθηκε κριτική από το ελεκτικό συνέδριο και έχει αλλάξει η δεύτερη παράγραφος. Έτσι τώρα ο χρηματοοικονομικός κανονισμό της ΕΠΟΛ που δέχτηκε κριτική από το ελεκτικό συνέδριο συνάδει με το δημοσιονομικό κανονισμό. Την τελευταία συνάντηση λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου το πράξαμε αυτό. Μας ρωτήσατε γιατί δεν υπήρξε βελτίωση νωρίτερα. Δεν μπορώ να σας δώσω μια σαφή απάντηση και ζητώ συγγνώμη. Γιατί η προηγούμενη δίκηση δεν έλαβε μέτρα νωρίτερα. Δεν έχουμε την πρόθεση, όπως σας είπα, να δικαιολογήσουμε ε, κανέναν για το τι έγινε στο παρελθόν. Θέλουμε όμως να βελτιώσουμε την κατάσταση το συντομότερο δυνατόν και με το βέλτιστο τρόπο. Έτσι λοιπόν, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν υπήρχε βελτίωση το 2008. Τώρα, για τις ε, ιδιωτικές δαπάνες και γιατί δεν έχει γίνει κάτι νωρίτερα σχετικά. Είχαμε μία σειρά ε, διαταγών ανάκτησης ε, έναντι κάποιων υπαλλήλων το 2008 και το 2009, αλλά δεν έχουμε καλύψει, δεν έχουμε ανακτήσει ακόμη το πλήρες ποσό τώρα. Έχει λάβει χώρα και ένας εξωτερικός έλεγχος ε, στον οργανισμό από, την εταιρεία, από μια εταιρεία μέτρα το Λονδίνο. Έχει υποβληθεί η έκθεση αυτή και στο λεκτικό συνέδριο και σε εμά. Ε, μία ακόμη συνέπεια αυτού του εξωτερικού ελέγχου ήταν ε, οι εντολέ ε, ανάκτηση που στάλησα στον πρώην διευθυντή, όπω σα ανέφερα. Ρωτήσατε για τις αλλαγές στον τομέα των προμηθειών, γιατί δεν έγινε αυτό νωρίτερα και τη βελτιώθηκε και από πού προέρχεται το εγχειρίδιο. αρμόδιος υπάλληλος ε, ε, ανέλαβε τα καθήκοντα το 2009 και το 2010 ε, μπόρεσε να βελτιώσει το σύστημα. Το εγχειρίδιο των προμηθειών βασίζεται σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, συλλέξαμε και όλες τις πληροφορίες και από τις άλλες υπηρεσίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Κυρία Ματιέ, ρωτήσατε για τις συναντήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι είχε αλλάξει σε σχέση με ε, το παρελθόν. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι εφαρμόσαμε ένα σύστημα υποβολής εκθέσεων και πάντοτε έχουμε πλήρη επισκόπηση του ε, προϋπολογισμού της χρηματοδότησης των προμηθειών σε κάθε τομέα έτσι ώστε η διοίκηση να έχει μια καλή εικόνα και να μπορεί να παρακολουθεί τι συμβαίνει στον οργανισμό. Επίσης από πέρσι έχουμε ένα audit panel που υποστηρίζει ε, το Διοικητικό Συμβούλιο. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε κάτι τέτοιο στον οργανισμό. Έχουμε ελεγκτές που έρχονται από τα κράτη-μέλη και ελέγχουν ε, το έργο του οργανισμού και υποστηρίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο και το βοηθούν να λάβει αποφάσεις αν υπάρχει κάποια σοβαρή παρατυπία ή κάποιο σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τη διαχείριση. Τώρα για τα σεμινάρια και τα μαθήματα. Να σας πω τι έχει αλλάξει. Δύο τι να θέλω να αναφέρω. Καταρχήν, από πέρσι αρχίσαμε να εφαρμόζουμε ένα σύστημα εταιρικών σχέσεων και συμφωνίων επιχορήγησης. Ε, δεν ε, ε, ε, τώρα ε, έχουμε αντικαταστήσει αυτές τις συμβάσεις με αυτές τις εταιρικέ σχέσεις πλαίσιο και βάσει αυτών υπογράφουμε τις επιχορηγήσεις για τις νέες δραστηριότητες. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε τις υπογραφές όταν θα έχουμε και το τεχνικό προϋπολογισμό. Θα μπορέσουμε να υπογράψουμε τότε και τις συμφωνίες επιχορήγησης. Αυτό ε, είναι το ένα και ο άλλος ε, τομέας ε, σημαντικός για τα κοινά προγράμματα είναι ο εξής. Έχουμε δεχτεί κάποια κριτική για αυτές τις συμβάσεις με τους εκπαιδευτές. Δεν υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις. Αλλάξαμε το σύστημα. Θα έχουμε μόνο ένα σύστημα συμφωνιών επιχορήγησης, όπως σας είπα, και είναι σε φάση ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Διαφορετικά, ευχαριστώ να σας δώσω περαιτέρω εξηγήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε να συζητήσουμε και σε εσά να δώσετε γραπτές απαντήσεις γιατί κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τα μέλη της Επιτροπής μας να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε μία ακόμη υπηρεσία, ένα ακόμη οργανισμό και δεν έχουμε χρόνο. Να ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν αν ικανοποιήθηκε με τις απαντήσεις της ΕΠΟΛ. Κομισιόν, μπορείτε να μας πείτε αν έχετε ικανοποιηθεί με τι απαντήσεις που δόθηκαν στο λεκτικό συνέδριο. Αλλά θέλω και να περάσω και στον τελευταίο οργανισμό, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Δύο κύριε ερωτήσεις έχω εδώ. Για την, τον οργανισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ένα έχει να κάνει με τις προσλήψεις και τις διαδικασίες πρόσληψης. τιμήσει ε, για σχέδια πρόσληψης ε, αν υπάρχουν σήμερα, σύμφωνα με τον οργανισμό. Και θέλω επίσης να θίξω και ένα συγκεκριμένο θέμα για ε, μια σύμβαση πλαίσιο που ε, δόθηκε για τέσσερα χρόνια τον Ιούλιο του 2007 αλλά μετά από δύο χρόνια και λιγότερο, η κονδύλια είχαν ήδη δαπανηθεί. Και δαπανήθηκαν περαιτέρω κονδύλια χωρίς περαιτέρω έγκριση από τον οργανισμό. Μπορεί να μα εξηγήσει λοιπόν ο οργανισμός ε, με σαφήνεια γιατί συνέβη κάτι τέτοιο. Να δώσουμε το λόγο καταρχήν στον εκπρόσωπο του οργανισμού και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν για να τοποθετηθεί για τις απαντήσει τη ΕΠΟΝ. Κύριος Μανολόπουλος, παρακαλώ. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Thank Ευχαριστώ, Πρόεδρε. με δύο ερωτήσει που είπαμε ο κ. Μπιζουτήλ. Καταρχήν, όσον αφορά τι εκτιμήσει προσλήψεων, θα ήθελα να σα διαβεβαιώσω ότι πήραμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιταχθούμε στις υπερβολικές εκτιμήσεις που κατέδειξε το ηλεκτρικό συνέδριο αυτό που θα να σας πω είναι ότι θα εισαγάγουμε μία νέα εκθέσεις για να μπορέσουμε να ελέγχουμε ακριβώς τι γίνεται όσον αφορά την εκτέλεση του προπολισμού για τον τίτλο 1. Δαφά πάνες λοιπόν για προσλήψεις. Αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι η δική μας υπηρεσία άρχισε να λειτουργεί το 2007 και περιμένουμε το 2008 για να γνωρίσουμε τον διευθυντή και αιτήσει της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ε, εμείς είχαμε δεχθεί να μην γίνει καμία πρόσληψη πριν να έρθει ο νέος διευθυντής. Και δεν μπορώ να σας σε αυτή τη στιγμή ότι πήρα τα αριθμητικά στοιχεία αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι έχουμε 50% ανοιχτών κενών θέσεων για το 2010. Πήραμε λοιπόν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε προγραμματισμό, έχουμε ένα ε, διευθυντή προγραμματισμού και τελικά θα έχουμε ένα πρόγραμμα με τέσσερις ε, προτεραιότητες. Προτεραιότητα 1, 2 και 3 και 4 και η 3 λέω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, της ανάλογης υπηρεσίας της Κομισιόν και αν έχουμε κάποιο πλεόνεσμα να το πω έτσι θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να πραγματοποιήσουμε ορισμένα από τα σχέδια που ζητάει το διοικητικό μας συνέδριο. Χωρίς να έχουμε εμείς τα χρήματα. έχουμε 99,4% στις ε, ε, υποχρεώσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία που λάβαμε την τελευταία εβδομάδα είδαμε το 2008 είχαμε διαγραφή πόρων 3% και το 2009 6% ε, από τα μεταφερθέντα ποσά και αυτό που είχαμε τελικά εκτέλεση πέρσι ήταν 98% που οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έχουμε δύο στόχους. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το, τη διαγραφή του 10% για τα μεταβερθέντα ποσά. Και το άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι δεν θα έχουμε κάτω από το 95% για τις ε, υποχρεώσεις. Το 2009 και το 2010 είχαμε 99,4 και το 2010 99,7 χρήσεις των πόρων μας. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν μεταφορές λόγω του τι κάνουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι εκθέσεις ε, που αναθέτουμε να πραγματοποιηθούν μέσα στα πλαίσια του ενός έτους. Ακόμα και αν ξεκινήσει δηλαδή η αίτηση υποβολής ε, προτάσεων τα αρχές του έτους θα μπορεί να υπάρχουν υπογραφές στη σύμβαση το Μάιο μετά πρέπει να συλλεχθούν τα στοιχεία υπάρχει πάντα μια καθυστέρηση γιατί ξεπερνάμε τα τέλη του έτους. <clears throat> Όσον αφορά τη συμφωνία πλαίσιο, ένα θέμα που έθεσε ο κ. Μπουζουτήλ για το 2007, αυτό είναι ε, μία σύμβαση πλαίσιο, δηλαδή πρόσληψης μιας εταιρείας για να οργανώνει διασκέψεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Το 2007 ε, δεν είχαμε το νέο διοικητικό συμβούλιο, δεν είχαμε το νέο διευθυντή. Όταν έφτασε ο νέος διευθυντής είχαμε μια διαφορετική μέθοδο λειτουργίας. Αποφασίσαμε από εκεί και πέρα να έχουμε μια ετήσια διάσκεψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγινε πριν από τα Χριστούγεννα εδώ στα, στις Βρυξέλλες που άλλαξε κάπως αυτή την ε, υποβολή προτάσεων που ήταν για 2 εκατομμύρια ευρώ στην αρχή, ευρώ στην αρχή και είχε ε, απορροφηθεί πολύ γρήγορα. Δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε πριν από την υπογραφή βέβαια της νέας σύμβασης και γι' αυτό το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε τελικά ήταν να ακυρώσουμε την αιτήσια αυτή διάσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε οργανώσει με την Σουηδική Προεδρία, κάναμε μια ανάλυση των κινδύνων και είπαμε ότι εντάξει θα συνεχίσουμε. Αλλά η σύμβαση ήταν νόμιμη και δεν λέει πουθενά το ηλεκτρικό συνέδριο ότι ήταν παράνομα αυτά που έγιναν μέσα στα πλαίσια αυτού του διαγωνισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας συνεχίσουμε εκτός αν έχει κανείς και άλλο ερώτημα, αλλά ας το κάνει γραπτός γραπτός. Όχι, εγώ θα προχωράσω στα συμπεράσματα μου, εκτός αν η Κομισιόν έχει να μας πει τίποτα. Α, πρέπει να μιλήσει και η Κομισιόν και μετά εσείς μετά. Η Κομισιόν λοιπόν, αλλά συντόμως για το πολύ εκεί πέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Κομισιόν θεωρεί ότι μετά την αλλαγή των πραγμάτων το ΣΥΠΟΛ άλλαξε πρόσωπο. Η νέα διαχείριση κάνει μεγάλες προσπάθειες για να βρει λύσεις στα εκκρεμή προβλήματα και η Κομισιόν υποστηρίζει τη λύση των προβλημάτων του ΣΥΠΟΛ ώστε να παραμείνει το κύριο εργαλείο για την εφαρμογή των στόχων της Στοκόλμης στην αστυνομική εκπαίδευση. Είχαμε ζητήσει να αλλάξει η διαχειρίση της υπηρεσίας αυτής και η Τσεχική Προεδρία το 9 τον Μάιο μάλιστα του 9 φτάσαμε στην αρχή του τέλους της θητείας του προηγουμένου διευθυντού. Ξέρω ότι το θέμα σας δεν είναι ο προπολογισμό του 9, αλλά καλό ήταν να το πούμε διότι το 2010 η υπηρεσία αυτή βελτίωσε πάρα πολύ τη χρήση του προπολογισμού της. Όπως είπε και το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο παράδειγμα. Τα ποσοστά το 10 δαπάνησε, απορρόφησε τέσσερις φορές περισσότερα ποσά από το 8. Ευχαριστώ. Ορίστε σύντομα συμπεράσματα και μετά θα προχωρήσουμε. Θα ζητήσουμε δε επέκταση τη χρόνου συνεδρίασης από τους διερμηνείς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα η γραμματεία να μας βοηθήσει εδώ Μας βοήθησαν και οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών και η ίδια η Κομισιόν, αλλά ό,τι κατάλαβα ενοχλήθηκαν και λίγο και για μένα ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζω να συμφωνούν όλοι ότι εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα διαφάνειας, διότι εδώ μιλάμε για χρήματα των φορολογουμένων και θα έπρεπε κάθε χρόνο να έρχονται να μας εξηγούν πώς δαπάνησαν τα χρήματα αυτά. Γιατί και εμείς με αυτή τη βάση θα δώσουμε την απαλλαγή. Επίσης χαίρομαι γιατί ο εισηγητής από την Κοκομπού, η Μόνικα Μακοβέη, παρίσταται και είμαι σίγουρος ότι θα το παρακολουθήσει το θέμα και για την γνωμοδότησή μας τον επόμενο μήνα ή μάλλον μέσα αυτό το μήνα. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Μπουζουτήλ θα υποβάλει επίσημα τη γνωμοδότησή του τη, στις 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου και η διορία κατά τροπολογιών λήγει την 5η 3 Φεβρουαρίου. Η δε ψηφοφορία στην ΕΛΕΦ θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή όλων και των εκπροσώπων των υπηρεσιών και θα θέλαμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις να τις απαντήσετε γραπητός. Έχουμε ακόμη ένα θέμα. Ακόμη ένα θέμα είναι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Φραζιλίας για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρηση βαρχία διαμονή για του κατόχου κοινών διαβατηρίων και διπλωματικών και άλλων. Συνεισηγητές είναι η Μόνικα Μακοβέη και ο Γιώαν Έντσιου. Παρακαλώ λάβετε το λόγο ταυτόχρονα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για το θέμα της κατάργησης των θεωρήσεων μεταξύ Ένωσης και Βραζιλίας συστήνω με βάση τις απόψεις του Κοινοβουλίου να εγκριθούν οι συμφωνίες αυτές και για τους Κυπρίους, Εσθονούς, Μαλτέζους κλπ. Να μην χρειάζεται βίζα για να μεταβούν οι κοινοτικοί αυτοί οι πολίτες εκεί είτε για δουλειά είτε για διασκέδαση. Οι Βραζιλιάνοι δεν χρειάζονται βίζα για διαμονή μέχρι τρεις μήνες αλλά για περαιτέρω χρειάζονται και οι κοινοτικοί ακόμη χρειάζονται θεώρηση για να μπουν στη Βραζιλία. Αυτό θα αλλάξει βέβαια. Θα ο Πάσα Ίσκ να πηγαίνει στη Βραζιλία χωρίς θεώρηση. Εφόσον λοιπόν υπάρξει συμφωνία του Κοινοβουλίου γενικότερα, συμφωνώ και εγώ. Και έπειτα ο κύριος Έντσου θα μας μιλήσει για τα διπλωματικά διαβατήρια. Ορίστε κύριε Έντσου για τα διπλωματικά. Ευχαριστώ. Θα θα ήθελα να συστήσω στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει αυτή τη συμφωνία. Οι διαπραγματεύσει γίνονται σε δύο φάσεις. Η συμφωνία για τα συνήθη διαβατήρια, για τα κοινά διαβατήρια, θα πρέπει να εγκριθεί από τα εθνικά κοινοβούλια, ίσω χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Υπάρχει όμω ξεχωριστή συμφωνία για τα διπλωματικά διαβατήρια αυτή η συμφωνία μπορεί αμέσως χωρί επικύρωση της Βουλής να τεθεί σε ισχύ εφόσον έχει προσυπογραφεί και εγκριθεί. Γι' αυτό υπήρχαν αυτές οι δι, διτές διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι για να μην χάσουμε χρόνο. να υπενθυμίσω στην Κομισιόν ότι έχει πραγματικά ε, αρμοδιότητες όσον αφορά τις εξωτερικές διαπραγματεύσεις για ε, τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Υπάρχουν ακόμα έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούν ακόμα να πάνε στην ΣΥΠΑ και στον Καναδά χωρίς ε, ε θεώρηση και θα ήθελα να τους ζητήσουμε να προετοιμάσουν παρόμοιες συμφωνίες για τις, τα κοινά διαβατήρια και για τα πραγματικά. Η Βραζιλία έδειξε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος. Δεν υπάρχει κανένα λόγο γιατί αυτοί που έχουν αυτά τα διπλωματικά διαβατήρια θα πρέπει να έχουν προβλήματα. Η Κομισιόν λοιπόν ήταν καλό να ξεκινήσει τι διαπραγματεύσει αυτέ με τι ΗΠΑ και τον Καναδά, του Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, η Τσεχία και η Κύπρος να μπορούν να διαταξιδεύουν χωρί διαβατήριο. Ευχαριστώ. Να ρωτήσω την Κομισιόν και την Προεδρία του Συμβουλίου αν θέλουν το λόγο. Παρακαλώ, Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω εκ μέρους της Κομισιόν να ευχαριστήσω τους δύο ε, για την ε, πλήρη υποστήριξή τους για αυτές τις συμφωνίες ε, απαλλαγής της θεώρησης με τη Βραζιλία και θέλω να σας ευχαριστήσω και για την πρόθεση επιτάχυνσης της διαδικασίας ε, προκειμένου να κυρωθούν αυτές οι συμφωνίες το συντομότερο. Και κάτι ακόμα, φυσικά η Κομισιόν θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες ε, για να διορθώσει τα υπόλοιπα προβλήματα που, που μένουν με την ε, ε, με τον Καναδά και τι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα και φυσικά θα λάβουμε υπόψη τι προτάσει που ακούστηκαν από το δεύτερο συγγητή. Ευχαριστώ. Άλλα σχόλια παρακαλώ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Επομένω, η προθεσμία είναι ε, την Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου, το μεσημέρι για τις τροπολογίες και 25-26 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί θα συζητηθεί, με συγχωρείτε, η γνωμοδότηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Σας ευχαριστώ. Πάνω κάτω, σεβαστήκαμε και το χρόνο, θα συνεδριάσουμε. Αύριο θα συζητήσουμε για... Μάλλον θα επιβεβαιώσουμε την έκτακτη συνάντηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τις 17 Ιανουαρίου, συνεδρίες συντονιστών, κατόπιν στις 25 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες και στις 26 Ιανουαρίου επίσης στις Βρυξέλλες θα συνεδριάσουμε. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Γεια σας. Exactly. <laughs> Thank you.